Καλημέρα σε όλους. Ε, πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρία... Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να σιγουρευτώ επειδή θα ψηφίσουμε ότι όλοι έχετε την κάρτα ψηφοφορίας και αν την έχετε ξεχάσει παρακαλώ στείλτε κάποιον να σας τη βρει, να σας την πάρει και να σας τη φέρει. Τι ωραία επιτροπή, πόσο πειθαρχημένη. Τέλεια, μπορούμε να αρχίσουμε. Σας υποβάλαμε το σχέδιο ημερησίας διατάξεως ήδη. Δεν πιστεύω να υπάρχουν αντιρρήσεις, ενστάσεις. Αν ε, δεν ε, ζητήσετε τροποποίηση ή υποβάλλετε ένσταση, θα εγκριθούν ε, στο τέλος της συνεδρίας τα πρακτικά όσα έχουν. Έχω την τιμή να αντικαθιστώ τον Μάλκολμ και θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Τι... Ο κύριος Κρόσμαν, τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, μία ανακοίνωση της Προεδρίας για να σας πω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίαση στο ίντερνετ. Καλώς ορίσατε λοιπόν οι θεατές μέσω ίντερνετ. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και έχετε αντιστοίχως τα έγγραφα στην είσοδο της αίθουσας. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε ως φίλοι της ΙΜΚΟ για να μπορείτε να λαμβάνετε και το ενημερωτικό φυλάδιο. Έχουμε τα πρακτικά της 10ης Ιανουαρίου, της 25ης, 26ης Ιανουαρίου και της 10ης Φεβρουαρίου που πρέπει να εγκρίνουμε. Μιλάμε για τις συλλογικές πρόσφυγες όπως επίσης και το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο, Α, δουλεύει, ωραία. Α, επίσης μέσα στο ενημερωτικό φυλάδιο θα, θα βρείτε και το τρίκ του μήνα. Και λέει πως μία επιχείρηση βγαίνοντας στο ίντερνετ μπορεί να υποφελείται και να επικαρπείται όλων των αγαθών της εσωτερικής αγοράς. Αυτόματα. Τα πρακτικά, πρακτικά δεν έχουμε, δεν έχουμε. Α, γυρνάμε σελίδα λοιπόν. Και πάμε στο πακέτο της σημερινής συνεδρίασης. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ θα μας μιλήσει για τη σύσταση της ονομασίας και της συναφούς επισήμανσης των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Ο κύριος Μάντερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Let me, uh, first... Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, για τη συνεργασία που είχαμε. Στην πρώτη ανάγνωση ε, εγκρίναμε τη 18η Μαΐου με μεγάλη πλειοψηφία τις υποβληθής ε, τροπολογίες με υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Πολλές τεχνικές τροπολογίες προφανώς αλλά και κάποιες ε, ουσιαστικές ή πολιτικές μπορώ να τις ε, χαρακτηρίσω. παραδείγματο χάρη η σήμαση περί προέλευση, ε, τα υποπροϊόντα, ζωικά υποπροϊόντα, ανεξάρτητα σήματα, ρήτρα αναθεώρηση κτλ. κτλ. Ε, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Υπουργική προεδρίας δεν μα είχε υποστηρίξει μέχρι τούδε. Τώρα σταδιακά αρχίζουν με την αλλαγή της Προεδρίας ε, να αποκτούμε μεγαλύτερη υποστήριξη. Λάβαμε και μια σχετική επιστολή και οι ενώσεις ε, θα υποστηρίξουν τροπολογία 4 σχετικά με τα προϊόντα και τα συστατικά ζωικής ε, προέλευσης. Άρα και το Συμβούλιο αποφάσισε να την προωθήσει αυτή την τροπολογία. Επίσης λάβαμε σήμερα μια επιστολή από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο υπέρ αυτής της τροπολογίας. Βήμα-βήμα λοιπόν σημειώνουμε πρόοδο. Κάνει κάποιους μικροφωνισμούς εδώ ο εξοπλισμός. Έχουμε λοιπόν, συνεχίζω, τις τεχνικές τροπολογίες ε, του Συμβουλίου, τις έχουμε γκρίνει στην πρώτη ανάγνωση, αλλά υπολείπονται, εκκρεμούν ακόμη κάποια ζητήματα. Επανησύγαγα κάποιες προτάσεις για διευκρινήσεις ε, ή απλουστεύσεις ε, ήδη εγκεκριμένων τροπολογιών. Μετά την πρώτη ανάγνωση λοιπόν. Φερρυπίν. η απέτηση αναφοράς ε, τη χώρα προέλευση των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων ε, με προέλευση τρίτη χώρα ε, βάσει και της πρότασης, αρχικής πρότασης του 2005 που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς το παρόν επ' αυτού δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο Συμβούλιο. Η τωρινή έλλειψη των ομοιόμορφων κανόνων σχετικά με τη σήμανση έχει ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρήσει τη να είναι σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με εταίρου από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, την Κίνα, την Ιαπωνία κτλ. κτλ διότι απαιτούν τη σήμανση προέλευση για τα εισαγόμενα προϊόντα. Και συζητήσαμε επίση με τι μεγάλε μάρκε εισαγωγικά, Nike, Adidas, Puma κτλ τους ε, παγκόσμιους αν θέλετε παίκτες, ε, τις ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα χρησιμοποιούν ήδη τη σήμανση προέλευσης διότι υποχρεούνται να αναφέρουν αυτή τη σήμανση στα προϊόντα, σου, προϊόντα τους συγγνώμη, για να τα θέσουν σε εμπορία στη ΣΥΠΑ παραδείγματος χάρη. Ε, ίσως λοιπόν βρούμε με κάποια λύση, προς το παρόν δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο Συμβούλιο. Επίσης, ε, Προ όφελο του καταναλωτή είναι να γνωρίζει που έχει παρασκευαστεί το κάθε προϊόν, αν έχει κατασκευαστεί ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές ε, τουλάχιστον γνωρίζουν ότι είναι κατασκευαστές, συμμορφώνονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ολόκληρο ο κόσμος ζητήσει, ε, την, ε, ζητάει μάλλον τη σήμανση προέλευση. το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς για να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ισότιμο ανταγωνισμό, ίσους όρους ανταγωνισμού και οι δικοί μας ε, κατασκευαστές για να ανταγωνιστούν τους υπολείπους στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης, η σήμανση προέλευση μπορεί να συμβάλλει ώστε να μειωθούν τα παραποιημένα προϊόντα ή την ψευδεπίγραφη δήλωση περί προελεύσεως Επίση, υπάρχει το εθελοντικό σύστημα σήμανση ε, της προέλευση ε, που μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν ε, υπάρχουν πολλές παραπλανητικές ε, πληροφορίες. Ε, βλέπουν οι καταναλωτέ ότι στο Βιετνάμ παραδείγματος χάρη έχει κατασκευαστεί ένα προϊόν, μετά στην επόμενη μπορεί σε ένα επόμενο στάδιο να έχει περάσει το προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γράφει μετά ότι κατασκευάστηκε στην Ολλανδία ή στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι παραπλανητική σήμανση και χρειαζόμαστε ε, ευκρινέστερες διατάξεις και για τις επιχειρήσεις ε, και για τους καταναλωτές ε, οπότε προτείνεται ως εθελούσιο αυτό το σύστημα σήμανσης. Αν κάνετε οπτήν, αν επιλέξετε να συμμετάσχετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αλλιώς δεν χρειάζεται να δηλώσετε ότι δεν συμμετέχετε στο σύστημα. τώρα τα κλωστοφαντουργικά προϊόντα ζωικής προελεύσεως ε, θέλουμε, επιθυμούμε μία απέτηση ε, που θα λέει ότι δεν υπάρχουν συνθετικά ζωικής προέλευσης μέσα σε ένα κλωστιφαντουργικό προϊόν. Προς το παρόν υπάρχουν γούνες και άλλα ζωικά υποπροϊόντα μέσα ε, σε κάποια κλωστιφαντουργικά προϊόντα. Οπότε οι καταναλωτές που δεν επιθυμούν να αγοράσουν ένα τέτοιο κλωστιφαντουργικό προϊόν θα πρέπει να έχουν τη σιγουριά και άρα θα πρέπει να αναφέρεται αν υπάρχουν δεν υπάρχουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. Διάκριση επίσης ανάμεσα στην πραγματική και την τεχνητή γούνα. Άλλο ένα θέμα. Είναι ε, δύσκολη διάκριση για τον... Ε, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση από τον καταναλωτή, να κρίνει ο καταναλωτής. Ε, πρέπει, επίσης, το ίδιο ισχύει και για το δέρμα. Πρέπει να αναφέρουμε αν είναι πραγματικό ή όχι το δέρμα. Προς το παρόν δεν προβλέπεται αυτό για τη γούνα, άρα θα χρειαστεί να αναβαθμίσουμε τις νομοθετικές διατάξεις και γι' αυτό. Προς το παρόν, ε, τα αυτορυθμιζό, το αυτορυθμιζόμενο και θελούσιο σύστημα ε, δείχνει, έχει καταδείξει ότι είναι ανεπαρκές και Και υπάρχουν πολλοί καταναλωτέ, παραδείγματο χάρη, που υποφέρουν ε, από κάποιε αλλεργίε και μπορεί να επηρεαστούν αν υπάρχει ε, ζωικό υποπροϊόν μέσα στο κλωστοβιοϊφαντουργικό προϊόν. Άρα ε, θα πρέπει να το γνωρίζει ο καταναλωτή να γνωρίζει τη σύνθεση του προϊόντο. Είμαστε ακόμη σε διαπραγματεύσει με την Ουγγρική Προεδρία για αυτό το θέμα και ελπίζω ότι θα βρούμε μια αποδεκτή λύση. Ε, ως προς τη ρήτρα αναθεώρησης, θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό ε, η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εγκρίνει πολλές προτάσεις, παραδείγματος χάρη. Μετά από την αξιολόγηση αντικτύπου ή τη διεξαγωγή μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρεπιπτόντως θα ρωτήσω την Επιτροπή αν έχει δρομολογήσει τη μελέτη, διότι πριν από ένα χρόνο μας είπε ότι με τα ε, θα ε, ζητήσει τη διεξαγωγή της μελέτης, μελέτης συγγνώμη, δεν ξέρω όμως αν έχει ξεκινήσει. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα, δεν υπάρχει καμία διαβούλευση για αυτό το ζήτημα, ίσως κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί μέσα στη μελέτη ζητάμε για τις αγορές ε, μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές ε, αν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί ένα ευρωπαϊκό μέγεθος για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, για την ένδυση κυρίως είναι εφικτό ή χρειάζονται άλλα εργαλεία σήμανσης ε, και όχι μόνο ε, ε, τη σήμανση που βλέπουμε πάνω στο προϊόν αλλά υπάρχουν άλλες πιο σύγχρονες μεθόδου, υπάρχουν πιο, πιο σύγχρονοι μέθοδοι που μπορούμε να εξετάσουμε να δούμε αν είναι εφικτό, αν είναι εύκολο να αντικατασταθεί το σύστημα να διερευνήσουμε ποιε είναι οι βέλτιστες ε, διαθέσιμες μέθοδοι ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτέ ε, και να διαπιστώσουμε αν μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, στο Συμβούλιο ζητήσαμε επίσης να υπάρχει σημάδι και για τις τεχνικές ίνες όχι φραστικά, αλλά για ένα παλτό ας πούμε ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ομοιόμορφο, μια ομοιόμορφη ευρωπαϊκή ή λατινική ονομασία. Ε, τώρα, ε, δεν είναι πρόσφορο να χρησιμοποιούμε πλέον 23 γλώσσες να αναφέρουμε σε 23 γλώσσες την κάθε πληροφορία και γι' αυτό προτείναμε να χρησιμοποιείτε μία μόνο ονομασία ή ένας κωδικός ή κάτι παρεμφερές. Αυτό θα το δει η αγορά. Αυτά θα προκύψουν από τη μελέτη και από τη διαβούλευση. Δηλαδή, οι αγορέ θέλουν να υιοθετήσουν αυτό το σύστημα και επίση είναι εφικτό ή μήπω συνεπάγεται υπερβολικό κόστο. Ε, επιθυμούμε την ε, ε, να λήξει η ρήτρα θεωρήσει μετά από 18 μήνες, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα, δυνάμει της ρήτρας αναθεώρησης, να προτείνει αλλαγές ανάλογα και με την ε, έκβαση, το πόρισμα της μελέτης. 18 μήνες ε, προτείνουμε ως χρονική περίοδο, ώστε να έχουμε χρόνο να προσθέσουμε, να προτείνουμε μάλλον κάποιες ε, βελτιώσεις για τον κανονισμό καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Ζητήσαμε λοιπόν και τους 18 μήνες, βλέπω τις σημειώσεις μου, τα έχω πει όλα αυτά. Α, επίσης, ε, βελτιώσαμε το κείμενο για τους απασχολούμενους ράφτες. Δεν χρειάζεται να ε, μπω σε λεπτομέρειες δεν εννοούσαμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, ε, δηλαδή ή αν στο διαδίκτυο ή αν στο ίδιο το κατάστημα μπορείτε να ζητήσετε εσείς ε, ε, κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μιλούμε για αυτές τις επιχειρήσεις, μιλούμε για τους αυτοαπασχολούμενους, για τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης για τα πειράματα στα εργαστήρια, για ε, τη σύνθεση των προϊόντων επιθυμούμε να εφαρμοστεί ε, το σύστημα της αμοιβαία αναγνώρισης. Δηλαδή αν έχει εγκριθεί κάποια ουσία, κάποιο συστατικό σε ένα εργαστήριο στην Ευρώπη θα θέλουμε να γίνεται αποδεκτό το πόρισμα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Ε, αφαιρέσαμε το κομμάτι για τα παιχνίδια δεν υπάρχουν πια διότι έχουμε τη σχετική οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών αλλά ε, πάντως για, τον, για τα πύληνα ε, ε, κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα με γούνα διατηρήθηκε η διάταξη. Θα περιμένω να ακούσω τώρα τους συναδέλφους μου. Εγώ δεν έχω άλλα εισαγωγικά σχόλια και θα επανέλθω στη συνέχεια. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κυρία Μάντες. Για όλες αυτές τις αναλυτικές πληροφορίες. Στην αίθουσα βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και του Συμβουλίου και στο τέλος της συζήτησης θα μιλήσουν. Τώρα, ο σκιώδης εισηγητής, η κυρία Κόμη απουσιάζει. Και είναι η κυρία Σαρτόρη που την αντικαθιστά. Κυρία Σαρτόρη, έχετε το λόγο. Μετά η Κριστέλ Σαρδεμοζέ. Για την Γκουε ποιος ε, θα πάρει το λόγο και ο Ματέο Σαλβίνη. Α, και αυτός λείπει. Ωραία, θα δούμε. Κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ εκπροσωπώ τη συνάδελφο Λάρα Κόμη, η οποία σήμερα απουσιάζει, διότι θα φτάσει αργά το βράδυ, δεν κατάφερε να είναι παρούσα. Η θέση που ψήφισε το Κοινοβούλιο στις 18 ε, του περασμένου Μαΐου είναι μια θέση που εκφράζει ευρέως ε, την πεποίθηση των πολιτικών ομάδων. Θεωρούμε όμως ότι οι τροπολογίες μας ε, ε, συνεισφέρουν στη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής που πρέπει να παλέψουμε για να περάσουν από το Συμβούλιο. Ο κανόνας της σήμανσης, της προέλευσης των προϊόντων που πρέπει να το παλέψουμε στη δεύτερη ανάγνωση, η ετικετοποίηση για τα υφαντουργικά από τρίτες χώρες και το προαιρετικό σήμα από τις χώρες της Ένωσης στοχεύουν σε δύο πράγματα. Ενισχύουν την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος αποκτά περισσότερη συνέστηση όταν αγοράζει, διότι ξέρει την προέλευση των προϊόντων του, και υποστηρίζει και τις επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες οι οποίες δεν έχουν ε, αλλάξει έδρα, δεν έχουν φύγει από την επικράτεια της Ένωσης. Δυστυχώς όμως η πρόταση του Συμβουλίου δεν έχει καμία αναφορά στην ονομασία προέλευσης. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Λιθουανία ζήτησαν την προαιρετική ονομασία προέλευσης. Αν το υποχρεωτικό σύστημα θεωρηθεί απαράδεκτο από το Συμβούλιο, Θυμηθείτε τι έγινε το 2005 όταν μπλοκάρισε για έξι χρόνια το Συμβούλιο την παλιά πρόταση και τώρα ξεκίνησε πάλι να προχωράει και αυτό λόγω της θέσης σε ισχύω την... της συναπόφασης και αυτό λόγω της κυρίας Μουσκαρδίνη και της δουλειάς της ε, στην Ίντα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τώρα πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να αξιολογήσουμε για ποιους λόγους υπάρχει αυτή η αντιμαχία και πρέπει να δούμε αν θα πρέπει, αν αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε για αυτούς τους λόγους την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεών μας. Ο κύριος Μάντερς θα πρέπει να συνεχίσει να υπεραμείνεται της ονομασίας προέλευσης. Για τα υπόλοιπα σημεία δεν έχουμε καμία άλλη διαφορά με τις θέσεις του εισηγητή. Ευχαριστώ. Η Κριστέλ Σαντεμόζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετική παρουσίαση αυτού του εγγράφου για τα κλωστεφαντουργικά. Θα είμαι σύντομη. Εγώ σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζω αυτά τα οποία υπόθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό όταν εργαζόμαστε για τις προτάσεις γύρω από τα κλωστεφαντουργικά να υπάρχει συνένεση στο Κοινοβούλιο για να μπορούμε μετά να είμαστε και ισχυροί στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους κλάδους, αλλά κυρίως για αυτόν εδώ τον τόσο σημαντικό κλάδο. Το θέμα της πληροφόρησης των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικό για μένα και η περίφημη ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση. Ο αυτό που, που είπε η Κομισιόν και το Συμβούλιο τι, είναι, ε, τι έχει ως στόχο είναι να προστατεύσουμε τους καταναλωτές που αγοράζουν κλωστιφαντουργικά προϊόντα. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει μία ρήτρα άμεσης παρέμβασης σε αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη σαφήνεια και τη συντομία. Η κυρία Άιντερχουλ για τους πρασίνους. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομα διότι χαίρομαι και προσβλέπω σε καλή επιτυχία με τις διαπραγματεύσεις και θα περιμένω να δω που θα καταλήξετε. Ακόμη πιο σύντομο και πιο σαφές. Οπότε επειδή ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά, τώρα θα αφήσω το λόγο στην κυρία Έμα Μακάρθη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αλλά έχω διάφορα να σας πω. Καταρχήν χαίρομαι ιδιαιτέρως για το σχέδιο της συστάσεως για δεύτερη ανάγνωση και για τις τροπολογίες του εισηγητή Μάντερς που προσπαθεί να απλοποιήσει το σύστημα και να επιτρέψει τις νέες σύνες στο ταχύτερο δυνατόν στην αγορά. Αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει και υποχρεωτική σήμανση προέλευση στην έκθεση αυτή και ε, να αναφέρεται το σύστημα και βεβαίως δεν συμφωνούμε με τα σύμβολα που βασίζονται σε γλωσσικές έννοιες διότι πιστεύω ότι ουσιαστικά αυτό θα περιέπλεκε την κατάσταση για τους καταναλωτές και θα πρέπει να είναι κάτι που θα λάβουμε υπόψη πριν την εφαρμογή. Απ' την άλλη πλευρά χαιρετίζουμε ε, την ε, είναι στάση σχετικά με την ρήτρα αναθεώρησης για τα αλλεργιογόνα διότι είναι κάτι που ανησυχεί τους καταναλωτές και θα πρέπει σαφώς να το αναφέρουμε. Κι εγώ όμως σας εύχομαι καλή επιτυχία για τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβόλαιο και περιμένω. Η Εύα Μπρίτ Σουίνσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Συμφωνώ με αυτό που ακούσαμε, ότι ουσιαστικά προσβλέπουμε στο να ακούσουμε τα σχόλια της Επιτροπής. Εμείς υποστηρίζουμε τις προτάσεις ε, του εισηγητή, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσω και τίποτα άλλο. Πλην δώσω το λόγο στην Κομισιόν, ποιος θέλει το λόγο. Η κυρία Ριγκογέν Πέρες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Ένα θέμα, ε, κάτι το οποίο λείπει και είναι ουσιαστικότατο για τον καταναλωτή και ο καταναλωτής όταν διαβάζει την ετικέτα και βλέπει τι σόι προϊόν θα καταναλώσει αυτό το οποίο κοιτάει πρώτα είναι το μέγεθος, το νούμερο. Λοιπόν δεν υπάρχει εναρμόνιση στα μεγέθη, στα νούμερα, πόσο στα ρούχα και στα παπούτσια. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μία εναρμόνιση των ε, μεγεθών για να μην ε, δημιουργούμε και προβλήματα δηλαδή στους νέους και στους λιγότερο νέους. Θα δώσω το λόγο τώρα γιατί είναι σημαντικό στην Κομισιόν, στον κύριο Λουίς Φιλίπε Ζιβάου και στη συνέχεια κόβεται το μικρόφωνο της Προέδρου στην κυρία Καταλίνα Γιακάμπα. Ο κύριος Λουίς Φιλίπε Ζεγάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε ήδη, σε προηγούμενες συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου και τις τροπολογίες που έχει βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδίως εφόσον αναφέρονται στη χώρα προελεύσεως και ε, ε, ε, τα υλικά πρέπει να πούμε ότι και στις δύο αυτές τροπολογίες όπως και σε άλλες νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει κάποια περαιτέρω επεξεργασία σχετικά με την διατύπωση των ε, τροπολογιών τεχνικά διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξουμε θεωρούμε ότι συνεχίζουμε να έχουμε δυσκολίες εις τον κανονισμό σχετικά με τα ανεξάρτητα σήματα, σύμβολα, δηλαδή θα πρέπει να το ξαναδούμε πριν εφαρμοστεί εις την στον ε, κανονισμό το θέμα των εργαστηρίων δεν έχει αναφερθεί ε, και θα θέλαμε να υπάρχει μία πιο σύντομη ρήτρα αναθεώρησης ε, για να έχουμε τη δυνατότητα να οργανωθούμε σχετικά με αυτό το θέμα. Τώρα υπάρχει μία νέα τροπολογία 12 με κάποια διατύπωση που προηγουμένως υπήρχε στην οδηγία και δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται στον κανονισμό απλώς θα πρέπει να λέγεται ότι τα προϊόντα πρέπει να συνάδουν με το, την νομοθεσία διότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει κάποια καθοδήγηση για την εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία και επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινάμε εργασίες για να προβούμε σε μία μελέτη για τις ε, άλλες δυνατότητες σημάνσεως των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων οπότε ακόμη και αν αυτά συνδέονται με τον κανονισμό παρόλα αυτά πιστεύω ότι ήδη θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την άσκηση θα προσπαθήσουμε να το ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν ταχύτερα. Δεν ξέρω εάν θα είναι 18-16 ε, ή πόσοι μήνες, αλλά θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση και εντός των επόμενων δύο ετών θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ε, μία αξιολόγηση τεχνική και οικονομική ε, και με τις τις νομοδοτήσεις των ενδιαφερομένων επί του θέματος. Θέλω να ολοκληρώσω με ένα άλλο θέμα που αναφέρεται στο θέμα των αλλεργιογόνων σε σχέση με τις ίνες. Και πάλι εμείς θα προτιμούσαμε αυτό να περιληφθεί στην αξιολόγηση και όχι στον κανονισμό, διότι δεν είναι ένα θέμα τεχνικό ή δεν είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι υπάρχουν αλλεργίες που συνδέονται με τις ίνες. Ουσιαστικά αναφέρονται εις τις χημικές και παρεμφερείς ουσίες, οπότε εάν εμείς κάνουμε αιτήσει από τις άμα, άμα επιβάλλουμε απαιτήσει θα πρέπει αυτό να περιληφθεί στον κανονισμό. Θα αφήσω τώρα το λόγο στην Ουγγρική Προεδρία την οποία ευχαριστώ για την Προεδρία της και την κυρία Καταλίνα Κάπατς ε, με συγχωρείτε για τον τρόπο που πρόφερα το όνομά της. Καταρχήν θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Μάντελς και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο σύστασης το οποίο και εξετάσαμε. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για τις εργασίες στην ομάδα εργασίας. Στις 25 Φεβρουαρίου την Παρασκευή είχαμε την πρώτη συνεδρίαση και για το θέμα της ονομασίας προέλευσης υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, ε, σοβαρές αντιρρήσεις από ορισμένα κράτη-μέλη. Ορισμένες άλλες, ε, για ορισμένες άλλες τροπολογίες ε, η στάση είναι πιο ελαστική. Θα προσπαθήσει η Ουγγρική Προεδρία να βρει έναν συμβιβασμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων και να προτείνει και να ολοκληρώσει μάλλον ε, την δουλειά μας, να τελειώσουμε τη δουλειά μας πριν από το τέλος της Προεδρίας. Η επόμενη συνεδρία είναι την επόμενη Παρασκευή. Θα δώσω το λόγο πολύ σύντομα στον κύριο Μάντερς πριν ε, σας ανακοινώσω ποια θα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ επειδή είχαμε ε, στενή και έχουμε στενή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές, ε, φαίνεται περιττό να μακρηγορώ εδώ. Δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Γιατί τους συναδέλφους που παρενέβησαν ε, σχετικά με τη σήμανση και τα σύμβολα ε, δεν γίνεται στα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, στα τρόφιμα, λέμε E71, ε, E363, ε, όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει το σύμβολο στα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα δεν ξέρω υποθέτουν ότι είναι αφελείς όσοι αγοράζουν κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα γιατί δεν χρειάζεται. Τώρα θα απαντήσω στον κύριο Ζεράρ για τις αλλεργιογόνες ουσίες. Χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται έρευνα νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα εξακριβώσω ότι έχουμε ήδη συμφωνήσει και, συμφωνήσει και θα επανέλθουμε. Η Δευτέρα Μαρτίου είναι καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και στις 21 Μαρτίου ε, ε, ε, εξέταση των τροπολογιών, την επόμενη μέρα ψηφοφορία και το Μάιο στην Ολομέλεια. Νομίζω έχουμε χρόνο για να λύσουμε τα προβλήματά μας που κυρίως θα έχουμε με το Συμβούλιο και σε πολύ μικρό το βαθμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μάντες. Εξοικονομούμε και χρόνο. Τετάρτη, 2 Μαρτίου μας είπατε, σε δύο μέρες δηλαδή είναι καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες, ε, μας είπατε όλες τι ημερομηνίε. Η απόφαση των συντονιστών σχετικά με την πιθανή έγκριση σε δεύτερη ανάγνωση έχει προβλεφθεί για τι 22 Μαρτίου. Η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για έγκριση με τη δεύτερη ανάγνωση, ε, αυτό τοποθετείται στην περίοδο ανάμεσα στο Μάρτιο και το Μάιο του 2011 και θα δούμε ε, αν θα ψηφίσουμε στι Μαΐου ανάλογα με την έκβαση του τριμερούς διαλόγου. Ε, ας περάσουμε τώρα στις τρεις επόμενες εκθέσεις ε, για την ενιαία αγορά. Θα τις πάρουμε έκθεση προς έκθεση για την ε, σαφήνεια της συζήτησης. Βέβαια συνδέονται στενά η μία έκθεση με την άλλη. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τη διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδους εισηγητές διότι εργαστήκαμε όντως σαν μία ομάδα και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους διότι συντονίσαμε τις εκθέσεις μας σε ορισμένα θέματα μεταξύ μας και για την διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση είχαμε 124 ε, ε, τροπολογίες, τις συζητήσαμε μεταξύ των τριών εισηγητών και συμφωνήσαμε ορισμένες από αυτές τις τροπολογίες οι οποίες είχαν υποβληθεί για τη μία έκθεση να, και ουσιαστικά αναφερόντουσαν σε κάποιο άλλο θέμα να μετατεθούν. Ουσιαστικά ε, προχωρήσαμε πολύ καλά με τους ε, ε, άλλους εισηγητές για να υπάρξουν συμβιβαστικές τροπολογίες και αυτές τις οποίες τώρα εξετάζουμε με συγχωρείτε κυρία Κανιούτε, όσοι βγαίνουν από την αίθουσα να βγαίνουν σιωπηλά και χωρίς φασαρίες, διότι είναι πολύ δύσκολο για την εισηγήτρια που προσπαθεί να παρουσιάσει το θέμα της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την επέμβασή σας. Αυτές λοιπόν οι συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες εξετάζονται τώρα αναφέρονται στα εξής θέματα. Πολιτική ηγεσία, το φόρουμ της ενιαίας αγοράς και 20 βασικά μελήματα, συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών, καλύτερη ε, νομοθετική ρύθμιση είναι και έξυπνη διακυβέρνηση, ε, να λύσουμε ορισμένα θέματα βάσει των κανονισμών για τις υπηρεσίες, να χρησιμοποιούμε κανονισμούς και όχι οδηγίες και να υπάρχει καλύτερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή. Κατά τρόπον ώστε στην επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο να καταλήξουμε όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες και να είναι έτοιμη η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στους κοιόδης εισηγητές, πρώτα στο Μήτρο Ρέπο. Εμείς ε, συνεργαστήκαμε πολύ θετικά με την κυρία Καλνούτε. Αλλά υπάρχουν ακόμη μερικά εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Για μας τους σοσιαλδημοκράτες μας ενδιαφέρει ο ανοιχτός διάλογος με την ε, κοινωνία των πολιτών και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι και το θέμα των συλλογικών δράσεων το συζητήσαμε όταν συζητήσαμε την έκθεσή σας πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα και το θέμα της πολιτικής ε, ηγεσία, της πολιτικής leadership είναι πολύ σημαντική. Υπό το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να, εργάζονται, να, να συνεργάζονται πιο στενά. Από διοικητικής πλευράς βέβαια αυτό το οποίο έχουμε είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ την εισηγήτρια όπως επίσης και την ομάδα των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Μόρτεν λέγει δεν είναι εδώ. Κάποιος από την Άλντε θα ήθελε το λόγο, όχι. Κυρία Αιντεχούλε. Ευχαριστώ. Έχουμε όντως συναντηθεί δύο φορές πολύ επικοδομητικά και πρέπει να πω στην εισηγήτρια και στους συναδέλφους της Γραμματείας ότι τους ευχαριστώ για την καλή συνεργασία Πιστεύω ότι μέχρι το Στρασβούργο θα έχουμε καταλήξει σε επικοδομητικούς συμβιβασμούς και θα αποσύρω τότε ορισμένες τροπολογίες υπέρ αυτών των συμβιβαστικών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσον αφορά τους άλλους συζητητές όντως η κατεύθυνση είναι η ίδια. Ευχαριστώ η κυρία Έμα Μακάρθη και εγώ Πρέπει να σας πω ότι είμαι σκιώδη στα περισσότερα θέματα σήμερα κυρία Πρόεδρε. Όντως η έκθεση είναι εξαιρετική και οι συμβιβαστικές ακόμη καλύτερες. Οπότε αναφερόμαστε ή στην ηγεσία ή στην ε, οικονομία της κοινωνικής αγοράς ή στην τροπολογία των πρασίνων που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση και θα ήθελα να σας πω ότι οι τροπολογίε μου 1 και 7 είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσουμε την καθημερινή πρακτική και συμφωνώ με τη ε, διατύπωση αυτών των συμβιβαστικών και πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερες, ε, ε, καλύτερους συμβιβασμούς, να έχουμε και μία αναφορά στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσουμε καλύτερες δεσμεύσεις του Συμβουλίου αλλά όλα αυτά θα σας τα υποβάλω και γραπτός. Όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες πρέπει να σας πω ότι δεν αλλάζουν πολύ την ουσία και τη μορφή του κειμένου αλλά θα πρέπει ίσως ε, όσον αφορά τη συλλογική επανόρθωση να ψηφίσουμε χωριστά. Στην ε, τελευταία συνεδρίαση που μιλήσαμε για το ADR θα και κάπου καταλήξαμε πιστεύω όμως ότι η κυρία Καλιέτε ε, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να συμβιβάσει τις διάφορες θέσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντογιόγκ δεν είναι εδώ γιατί γκουε μήπως ο κύριος Τριανταφυλλίδης θέλει κάτι να σχολιάσει. Θα πω κάτι την επόμενη, στο επόμενο θέμα που είμαι ισχυώδης εισηγητής. Εντάξει. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε λοιπόν τρεις εκθέσεις σχετικά με την ε, πράξη ενιαίας αγοράς. Εφόσον λοιπόν το χρονοδιάγραμμα είναι το ίδιο και η Επιτροπή εξετάζει και τις ε, τρεις εκθέσεις, ε, το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να ανακοινωθεί στο τέλος των τριών εκθέσεων και να υπάρξει μια συνθετική αντιμετώπιση όλων μαζί. Εάν λοιπόν συμφωνείτε, τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη έκθεση για την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Αντώνιο Φερνάντο Κορέοντε Ντεπάντκάντπος. Ευχαριστώ πολύ. «276 τροπολογίες λάβαμε και οι 52 από αυτές αφορούν στο κεφάλαιο περί προτεραιοτήτων. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη διάσταση απόψεων. Έχουμε ε, κάνει διάφορες συναντήσεις ε, με τους σκιώδεις συζητητές... Συναντήθηκα, διορθώνει ο με ε, τους ε, σκιώδεις και τους λοιπούς εισηγητέ, ε, των άλλων θεμάτων δηλαδή. Είχαμε αγαστή συνεργασία και στις μεν και στις δε. Ε, στις 16 Φεβρουαρίου συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές και είπαμε θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ενιαία συμβαστική λύση για τις προτεραιότητες, ούτως ώστε να είναι ισχυρή και συνενετική η τελική μας θέση το θέμα των προτεραιοτήτων και της θέσης, της ισχύω αν θέλετε, αυτής της οδηγίας είναι συνάρτηση της ικανότητας του Κοινοβουλίου να μιλήσει με μία φωνή και να μην φανεί η διχογνωμία για το θέμα αυτό. που σχετίζεται με την έκθεση Γκρέκ και την έκθεση του ε, κυρίου Μάριο Μόντι όπου φαίνονται ε, οι πλέον ρηξικέλευτε διαστάσει ε, του εγχειρήματο αυτού τη τόνωση δηλαδή τη ενιαία αγορά, ούτω ώστε να εξέλθουμε πιο αποτελεσματικά και από την κρίση ε, αποσκοπούμε σε μια ενιαία θέση όπως σας είπα επιθυμούμε να συνδράμουμε τον επίτροπο Μπαρνιέ στις προσπάθειες που κάνει για την πράξη της ενιαίας αγοράς. Πληθώρα θεμάτων λοιπόν που καλύπτουμε σε αυτές ε, τις τρεις εκθέσεις. Όπως ακούσαμε ήδη έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος. Ε, κρίνω πως ε, υπάρχει συμφωνία για βασικά ζητήματα παραδόξως πως ε, κανένας ε, δεν έχει ε, σημαντικές δαφικές αξιώσεις αν θέλετε. Δηλαδή όλοι κινούνται μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σήμερα μοιράσαμε στους κοιόδης εισηγητές και στους εισηγητές των λοιπόν εκθέσεων τις επτά προτεραιότητες Προτείνει ο εισηγητή 7 προτεραιότητε. Πρώτον, αμοιβή αναγνώριση δεξιοτήτων και ευρωπαϊκό διαβατήριο ικανοτήτων. Κατόπιν, ασφάλεια των ε, προϊόντων και έλεγχο εποπτεία των αγορών. Τρίτον, ε, βασικέ τραπεζικέ υπηρεσίε. Συγκρισιμότητα ε, των τελών και ενοποιημένη προσέγγιση. Τέταρτη προτεραιότητα που συνδέεται με την κινητικότητα των εργαζομένων και με τα δυνατότητα μεταφορά των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων δικαιωμάτων. Πέμπτον, ενιαία κοινωνική ρήτρα σε όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζεται με την ενιαία αγορά. Έκτη προτεραιότητα ε, και Κατάργηση των, ε, των τελών ε, roaming μέχρι τον 2012 και κατόπιν υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω και δεν είναι επίσημο γιατί δεν ήμουν επικεφαλής της αποστολής αλλά την περασμένη εβδομάδα διάφοροι ήμασταν ε, ε, στην Ουγγαρία στην επίσκεψη της Επιτροπής ΥΜΚΟ και συναντηθήκαμε με Ούγγρους βουλευτές της ομότυπης Επιτροπής του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας και συζητήσαμε κυρίως για την πρώτη και τη δεύτερη προτεραιότητα Δηλαδή, επιμείναμε στην αναγκαιότητα, αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου, καθώς και για το θέμα τη ασφάλεια ε, των προϊόντων. Ε, έχουν αναδειχθεί σε βασικές αυτές οι δύο προτεραιότητες ε, και ήθελα να σας τονίσω και πάλι ότι σας ενημερώνω προσωπικά. Δεν είναι η επίσημη ενημέρωση μετά από την αποστολή, σε καμία περίπτωση αυτό που ακούσατε. Όπως σας είπα, ε, θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις. Κατά πάσα πιθανότητα αύριο ε, θα κοινοποιήσουμε τις συμβαστικές λύσεις ε, για τις συμβαστικές τροπολογίες από των οποίων εργαζόμαστε. Και σήμερα ακόμη, αν είναι δυνατόν, Εφόσον ε, έλαβαν ε, ισχυώδεις εισηγητές πριν από δύο-δυόμιση ώρες, ε, εφόσον έλαβαν λοιπόν το έγγραφο με τις προτάσεις που συνιστούν για μας προτεραιότητα, αν τυχόν έχουν τώρα προτάσεις ισχυώδεις εισηγητές, με χαρά ήδη σήμερα να τις ακούσω. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πνεύμα συνεργασίας που δείξατε καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και διαβουλεύσεών μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Βαντούν δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σουάμπ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την έκθεση του εισηγητή Κορέαντε Κάμπους διότι την περασμένη εβδομάδα ε, θίξαμε ορισμένα θέματα όταν συναντηθήκαμε και για την σκιώδη συγγήτρια την συνάδελφο Φοντούν πρέπει να πω ότι ε, υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία δεν συμφωνεί ε, με τον εισηγητή υπήρξαν πολλές τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες αλλά Θεωρούμε θετικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμβιβαστικές τροπολογίες για τα ε, θέματα κλειδιά και θεωρώ ότι είναι θετικό και έτσι αντιμετωπίζει και η κυρία Τούν ότι διαγράφεται μία διέξοδος για συμβιβαστικές λύσεις αλλά οι τροπολογίες του συναδέλφου Κορέας Δικάμπος αναφέρονται μόνο στις προτεραιότητες και παραμένουν ακόμη σε κρεμότικα πολλά θέματα που ενδιαφέρουν την ε, ε, ομάδα του ΕΛΚ ε, και πέραν του ΕΛΚ ε, ορισμένες ε, επιφυλάξεις και των φιλελευθέρων και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι κοινωνικές επιπτώσεις διότι έτσι όπως προτείνει ο εισηγητής δεν επιτυγχάνει κανείς ούτε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα ούτε είναι εφικτή η λύση και θέλουμε να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε προτείνει διάφορες λύσεις από πλευράς ΕΡΚ για τη μείωση των τελών, για μία ενιαία αντιμετώπιση των ε, ε, επαγγελματικών ε, τίτλων και για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κατά τρόπεν αφενός για να υπάρχει μια ενιαία αγορά αλλά να μην καταστρέφονται και τα κίνητρα για τους εργαζομένους και γι' αυτό πιστεύουμε ότι τελικά πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες αυτό που αναμένουν από μας να παραμείνουμε και να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση και αυτό θα είναι ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω καταρχήν ότι η έκθεση, ε, η συζήτηση την οποία κάναμε με ε, τον εισηγητή στο Στρασβούργο ήταν πολύ επικοδομητική, προχωρήσαμε αρκετά και καταρχήν βλέπουμε ε, σύντομα επειδή υπάρχει στενό της χρόνου ότι και οι συμβιβαστικές λύσεις δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα προκύπτει όπως είπε ο συνάδελφος Σβάμπ ότι είναι η κοινωνική ρήτρα που πάντοτε ενδιαφέρει τους σοσιαλδημοκράτες αλλά πρέπει να δούμε αν δεν μπορεί να είναι πιο ευρία αυτή η διατύπωση διότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ε, μόνο τις επιπτώσεις της περιβαλλοντολογικές αλλά και τις επιπτώσεις στην απασχόληση και να δούμε ε, τι μπορεί να είναι και οι επιπτώσεις στον κοινωνικό χώρο γιατί θα, θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ίσως από αυτά τα οποία ζητούν οι σοσιαλδημοκράτες γιατί ε, θα πρέπει η ρήτρα αυτή να είναι πιο κοινωνική. Αλλά όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούμε να κάνουμε μία λύση one size fits all διότι υπάρχουν διαφορετικές δομές στα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα ήταν καλύτερα για να επιτύχουμε καλύτερα το στόχο μας να επεμβαίνουμε σε συγκεκριμένα σημεία, να μην προσπαθούμε συλλήβδη να λύσουμε τα πάντα και ακόμη και εδώ είναι προφανές ότι η οδηγία έχει ένα πυρήνα ελαχίστων κοινωνικών προδιαγραφών αλλά χρειάζεται και ευελιξία και ιδίως ε, να ληφθούν υπόψη τα, οι εθνικές ε, ιδιομορφίες, τα διαφορετικά κοινωνικά συστήματα διότι ε, λέμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμφωνούν επί των μισθών και ημερομισθείων και δεν μπορούμε εμείς από εδώ να λύσουμε όλα τα προβλήματα της Ευρώπης αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε με τον εισηγητή να δούμε ε, τις συμβιβαστικές προτάσεις που έχει κάνει για να έχουμε μία ενιαία αποδεκτή λύση διότι τότε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το Single Market Act και να του δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ σε όσους θέλουν να μιλήσουν να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας ε, πριν συναντήσουμε τους συμβιβασμούς που μπορούν να ικανοποιήσουν όλους κυρία Τσχούνεν δεν είναι εδώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί δεν έχω δει αυτόν τον ενημερωμένο κατάλογο των προτεραιοτήτων αλλά θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή διότι θεωρώ ότι η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες είναι βασικό αλλά αυτός ανεφέρθη γενικότερα στην ενιαία αγορά και εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι αναφερόμαστε ε, στην αγορά δανεισμού για τους καταναλωτές και χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε responsible lending και την τελευταία φορά δεν ήταν σαφής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε και έχω μία ερώτηση και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό ότι οι φιλελεύθεροι πρότειναν το θέμα της υποχρεωτικής κοινωνικής μελέτης των επιπτώσεων η οποία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να είναι πιο συγκεκριμένη και να γνωρίζουμε επακριβώς τι εξετάζει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακλάρκιν, πολύ σύντομα. Μιλώ εξ ονόματος του Μάλκομ Χάρμπορ, του πρόεδρου μας. Υποστηρίζει ο Μάλκομ τη σκληρή εργασία του κυρίου Κορέι Αντεκάμπος για αυτό το θέμα και να περάσετε ως πρακτικές παρατηρήσεις. Περιμένει το συντομότερο δυνατόν τις τροπολογίες. Ε, σήμερα το απόγευμα ε, θα ήταν το ιδανικό και ε, μετά στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα μπορεί να γίνει κάποια έκτακτη συνάντηση για να δούμε αν είναι εφικτό το σχέδιό μας. Ε, συνεχίζει τις προσπάθειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ καλωσορίζει τις καινοτόμες προτάσεις της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και από αυτόν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τώρα, για τις προτεραιότητες τις λάβαμε σήμερα το απόγευμα. Με την τωρινή διατύπωση, οι τροπολογίες 4 και 5 θα μας δημιουργήσουν κατά πάσα πιθανότητα ε, προβλήματα. Αντίθετα μπορούμε να υποστηρίξουμε τις 3 και 7 ε, στην επόμενη συνάντηση με τους Σκιώδης και με τον εισηγητή φυσικά θα συζητηθούν ε, όλα αυτά. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία, δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο και ελπίζω να με συγχωρήσει ο Μάλκομ γιατί τα είπα και πολύ γρήγορα και πολύ συνθετικά. Ευχαριστούμε. Κύριο Τριανταφύλλης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον, τον εισηγητή. Να πω ότι εμείς ε, συμφωνούμε με την προσέγγιση του η οποία καθιερώνει ως πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική διάσταση και που γενικά υποδεικνύει ότι η νέα ατζέντα για την ενιαία αναγορά πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε ωστόσο καταθέσει μια σειρά από ε, τροπολογίες που ε, εξυπηρετούν τρεις στόχους. Πρώτη λέμε να τεθούν ποσοτικοί στόχοι για την αξιολόγηση της εσωτερικής αγοράς βασιζόμενη σε κοινωνικά πρότυπα. Δεύτερον, οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια ή γενικού οικονομικού ενδιαφέροντο πιστεύουμε δεν πρέπει να καλύπτονται από το δίκαιο περί ανταγωνιστικότητα ή την νομοθεσία τη ενιαία αγορά. Και τρίτον, να ληφθεί υπόψη η συμβολή των κοινωνικών φορέων στη διαβούλευση για την ενιαία αγορά. Αυτά και θα συνεχίσουμε στι επόμενε συναντήσει με τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci. Je vais maintenant laisser la parole. Η κυρία Γκέπχαρτ. Αλλά Εβελίν, σε κοίταζα και φαντάζομαι ότι θα ήθελες να πεις τα ίδια πράγματα με μένα, οπότε δεν παίρνω εγώ το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Μπερναντέτ. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ αμφιλεγόμενο και με ενδιαφέρει είναι η κοινωνική ρήτρα διότι νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρανόηση στη συζήτηση για το τι συζητάμε όταν σαν σοσιαλδημοκράτες απαιτούμε αυτή τη κοινωνική ρήτρα διότι λέμε ότι είναι απαραίτητο αυτό το οποίο προβλέπεται στις συνθήκες επανελήφθη στη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή κοινωνική ε, ε, οικονομία αγοράς και οι άλλες ρήτρε οι οποίες υπάρχουν όντως να υλοποιηθούν και να, λέμε, και να διακηρύσουμε σαφώς ότι αυτό το κοινωνικό στοιχείο πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν είναι κάτι το αφηρημένο διότι μια τέτοια ρήτρα υπάρχει και στην ε, ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Ίσως λοιπόν πρέπει να τη ξανακοιτάξετε αυτή την οδηγία για να δείτε ότι το δικαίωμα το οποίο προβλέπεται σε αυτή την οδηγία δεν βλάπτει καθόλου καθόλου το δικαίωμα εργασίας ε, στη, στα κράτη-μέλη. Απλούστατα ε, αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και τίποτα παραπάνω. Όταν όμως μιλάμε ε, στο ΕΛΚ και στους φιλελεύθερους για κοινωνική ρήτρα και αν αυτό προβληματίζει αυτές τις δύο πολιτικές ομάδες τότε ο συνάδελφός μας Κορέοντε Κάμπος ίσως θα σκεφτεί μήπως μπορεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη έννοια αλλά πιστεύω ότι αυτή η νέα όθηση η οποία υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να χρησιμοποιηθεί διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει στο να δεχθούν αυτές τις προβλέψεις οι πολίτες της Ευρώπης. Ε, αντιθέτως η αξιολόγηση είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή πρέπει να αξιολογήσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε και εκεί χαίρομαι διότι οι φιλελεύθεροι μας είπαν ότι ευχαρίστως θα συζητήσουν το θέμα μαζί μας γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Βάιλερ. Κύριε Κρόιτσμαν, σε εσά απευθύνομαι, διότι πριν από ένα μήνα περίπου παρουσιάσαμε τη γνωμοδότησή μας για τη νέα μορφή του impact assessment, δηλαδή της αξιολόγησης των επιπτώσεων. Και εκεί είχαμε μία μικρή πλειοψηφία για impact assessment που στο τέλος θα εξετάζει και τις καταναλωτικές επιπτώσεις και ε, τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα και πολύ σωστά Βεβαίω ε, σκεφτείτε πού θέλετε να καταλήξετε διότι πολύ σωστά είπατε ότι στη Γερμανία και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη οι ε, συμβαλόμενοι κοινωνικοί εταιροί είναι ε, δεσμευμένοι από τις συλλογικέ συμβάσεις. Αλλού όμως οι διατάξεις καθορίζονται από το κράτος. Παραδείγματο χάρη για το δίκαιο εργασία. στη Γερμανία αυτό καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους ή οι λογικές συμβάσεις. Ε, υπάρχουν δηλαδή πάντοτε τομείς ασχέτως από τους μισθούς, ακόμη και το ημερομίσθιο εξαιρείται, που είναι όλοι αυτοί οι τομείς που δεν ρυθμίζονται μόνο από τους κοινωνικούς εταίρους παρόλο που για τα άλλα θέματα ε, πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Ε, ευχαριστώ. Κανένας άλλος δεν ζήτησε το λόγο. Πάμε τώρα στο τμήμα επιχειρήσεις και ανάπτυξη. Ο κύριος Μπουσόη έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας, δηλαδή τις τροπολογίες που υποβάλλετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για την Επιτροπή μας. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες και επεξεργαζόμαστε τις συμβαστικές τροπολογίες τώρα. Δεν πρόκειται μόνο για αυτή την έκθεση, δεν είναι δική μου η έκθεση. Εξάλλου είναι η έκθεση της Επιτροπής και ο στόχος να οικοδομηθεί μια ε, συμβαστική λύση για να τύχει υποστήριξη η έκθεση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Προφανώς η πληθώρα των τροπολογιών αντισχεραίνουν το έργο μας, δείχνουν μεγάλη διάσταση απόψεων. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να υιοθετηθούν ε, οι περισσότερε δυνατέ τροπολογίε. Έχω κυκλοφορήσει 16 συμβαστικέ ε, τροπολογίε ε, ε, που καλύπτουν τι περισσότερε τροπολογίε. Ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, πνευματικά δικαιώματα, άρνηση, όρια ανταγωνισμού, αθέμητο ανταγωνισμό ε, και ούτω καθεξή. Είναι θέματα που καλύπτονται από αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Θα ήθελα να κάνω και κάποιε παρατηρήσει για να κατανοήσετε γιατί δεν συμπεριέλαβα κάποιε τροπολογίε μέσα στι συμβαστικέ και γιατί συμπεριέλαβα κάποιε άλλε. Η αρχική τροπολογία μπορεί να αφορούσε σε μια διαφορετική παράγραφο, παραδείγματο χάρη. Ποιο είναι ο στόχο τη έκθεση, ε, να ιεραρχήσουμε τα μέτρα που θεωρούνται ω πλέον σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό επιμένω να έχουμε μία μόνο παράγραφο με στην έκθεση για κάθε επιμέρους θέμα. Αν ε, παραταθεί το κομμάτι που αφιερώνουμε σε κάθε θέμα δεν θα είναι αποτελεσματική η έκθεση. Θέλω να είναι συνθετική στο μέτρο του δυνατού και γι' αυτό στις προτάσεις μου συμβαστικές τροπολογίες που υπέβαλα έχω συγχωνεύσει τις παραγράφους που φέρουν επί του ίδιου θέματος και τις ε, τροπολογίες ε, που φέρουν επί του ίδιου θέματος. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να βασιστούμε μόνο σε προηγούμενη εργασία αλλά να βασιστούμε σε αυτέ τι προτεραιότητε που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή του και επίση να προαγάγουμε δικέ μα καινοτόμε ιδέε και ιδέε άλλων που μα ικανοποιούν. Στο Στρασβούργο την Τετάρτη σε 9 Μαρτίου θέλω να συναντηθώ με του ε, σκιώδει ηγητέ για να συντονιστούμε πριν από την ψηφοφορία. Ε, Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, θα σα πω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία για το συντονισμό τριών εκθέσεων και γνωρίζω ότι ε, θα συζητήσουμε στο Στρασβού αν τελικά θα καταθέσουμε κοινό ψήφισμα ή όχι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας δεν είναι εδώ. Για το ΕΛΚ θέλει κανείς το λόγο. Στη θέση του κυρίου Κάρας. Όχι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Κρίστιαν Μπουσόη για τη δουλειά του, για τη συλλογική δουλειά συνεργαστήκαμε όλοι αρμονικά για τις 16 συμβιβαστικές προτάσεις Πιστεύω ότι όλες διέπονται από τον κοινό νου. Τις έλαβα βέβαια αργά και στα αγγλικά, οπότε δεν μπόρεσα να τις εξετάσω. Θεωρώ ότι σίγουρα θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Υπάρχει όμως ένα σημείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε στις 9 Μαρτίου. Πρόκειται για το θέμα των καθολικών υπηρεσιών. Η γαλλική αντιπροσωπεία πραγματικά καίγεται με αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που ε, είναι εγκάσιο και στις τρεις εκθέσεις, ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ε, καταναλωτές, αποτέλεσε και ήδη έπαιξε σημαντικό ρόλο ως αμορτισέρ της ε, κρίσης αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και για τις ε, επιχειρήσεις και γενικότερα για την κοινωνία. Για τις ε, δημοπρασίες και τους διαγωνισμούς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία με τους ιδιώτες ε, με τις επιχειρήσεις, ε, ξέρουμε ότι το κράτος ε, δεν έχει πια και τόσους πόρους και αυτή η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να δούμε δηλαδή τι λειτουργήσε μέχρι τώρα σωστά, τι δεν λειτουργήσε για τις υπηρεσίες, η προσέγγιση σας είναι θετική σίγουρα, αλλά πρέπει να δούμε πού δούλεψαν τα πράγματα, πού λειτουργήσαν και σε ποιες χώρες δεν λειτουργήσαν καθόλου. Τελευταίο τώρα για τις προτεραιότητες τις οποίες μπορούμε να αντισταθμίσουμε φαντάζομαι και να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Συσπυρώνοντας και όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές ομάδες γύρω από την έκθεση Το πλαίσιο που προτείνετε δεν με ενδιαφέρει, δεν το βρήκα και τόσο ενδιαφέρον. Βρήκα όμως την εξαγγελία των προτάσεων πολύ σημαντική και η τροπολογία 38 που υπογράψαμε η Βελίν Γκεμπάρ και εγώ ε, είναι μια τροπολογία που ήδη έχει περάσει με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα στο πλαίσιο της έκθεσης της Περβάνς ε, Περέζα. Παρακαλώ την επόμενη εβδομάδα και εσείς να είστε ε, συνεπείς με αυτό το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί στην Ολομέλεια. είναι πολύ καλό ότι τώρα μιλάω μετά από την κυρία Βερνιό διότι πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην συμβάλλουμε στο να υπάρχει κατακαιρματισμός της νομοθεσίας και εδώ αναφέρουμε στις ε, παραχωρήσεις ε, σχετικά με τις, ε, την οδηγία των υπηρεσιών στην πράσινη βίβλο διότι έχει αναλυθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μια αναθεώρηση του θέματος. Για να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει απλοποίηση σε αυτό το θέμα δεν έχει σημασία αν ένα ή δύο μήνες ε, πριν υπάρξει μια χωριστή νομοθεσία που να αναφέρεται στα ίδια θέματα της οδηγίας των υπηρεσιών διότι έτσι υπάρχει κατακαιρματισμός γίνεται περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσουμε από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, καθορίσει ένα ενιαίο πλαίσιο και να μας κάνει μία ενιαία πρόταση και όχι ε, κατακαιρματισμένα προτάσεις θέμα. και σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Βελνιό για τις συνεργασίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα υπάρχουν νέα προγράμματα και εδώ δεν πρέπει να εφεύρει την πυρίτιδα το Συμβούλιο αλλά να κοιτάξουμε πώς θα υπάρξουν κοινά προγράμματα όπως έχει προτείνει και ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ. Σήμερα ε, μιλώ για τον κύριο Κουζούσνικ σχετικά με την έκθεση Μπουσόη και συμφωνούμε ότι είναι πολύ καλή και γι' αυτό δεν υποβάλαμε και τόσες τροπολογίες. Στηρίζουμε λοιπόν τις ε, τις κινήσεις σας για να υπάρξουν σωστές τροπολογίες στην πράξη ενιαίας αγοράς για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις αλλά εγώ θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα που θεωρεί πολύ βασικά η τροπολογία 5 του ηλεκτρονικού εμπορίου η τροπολογία 7 η οποία υποτίθεται ότι είναι συμβιβαστική ενώ μιλάει για εναρμόνιση του συμβατικού δικαίου και δεν ξέρω αν μπορούμε να δεχθούμε σε αυτή τη στιγμή διότι ακόμη γίνονται διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραμένουμε και την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το συμβατικό δίκαιο. Οπότε ε, το εταιρικό δίκαιο. Οπότε υπάρχει επίσης και ένα άλλο θέμα ε, όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει αποδυνάμωση των θέσεών μας ε, και στην τροπολογία 124. Στην τροπολογία τροπολογία 113 για την ενιαία φορολογική βάση ε, πιστεύω ότι η τροπολογία Edwards δεν έχει περιληφθεί στο σημείο αυτό ενώ θα έπρεπε να έχει παρατεθεί και παρακαλούμε να την λάβετε υπόψη σας. Η τροπολογία 16 για τις υποχωρήσεις στις υπηρεσίες ε, δεν συνάδει με την πρόταση Κουζούσνικ αυτή τη στιγμή και πρέπει να διατηρήσουμε τις προτεραιότητες της ενιαίας αγοράς. Πρέπει λοιπόν όπου είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις τροπολογίες ε, τις προτεραιότητες τις οποίες ήδη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις ανταλλάξουμε νέες ε, προτεραιότητες. Η κυρία Σβένσον. Ευχαριστώ πρόεδρε και χίλια ευχαριστώ προς τον κύριο Μπουσά και να ευχαριστήσω και τους άλλους δύο εισηγητές ε, παρεπιπτόντος γιατί με ρημνούν ώστε οι τροπολογίες που καταθέτουμε να ε, καταλήγουν στο σωστό σημείο, ας το θέσω έτσι. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μία προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για την κοινωνική ρήτρα, την κοινωνική διάσταση και ούτω καθεξής. Ακόμη και για αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με την ανάπτυξη και το επιχειρηματοϊκό πνεύμα θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της κοινωνικής ρήτρας. Ακόμη για τις επιχειρήσεις, ακόμη και για την ανάπτυξη είναι σημαντικό να τονιστεί αυτή η διάσταση δεν είναι ε, ε, οι τίτλοι σημαντικοί. Σημαντική είναι το περιεχόμενο και οι επιπτώσεις των μέτρων που θεσπίζουμε. Θα ήθελα τώρα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ε, σημασία των διασυνοριακών ε, συναλλαγών και τη σημασία που έχουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην ομάδα μας έχουμε υποβάλει τροπολογίες που σκοπό έχουν να τονίσουν έτσι ναι, περαιτέρω τη βαρύτητα του δημοσίου τομέα ακόμη και για τις, ε, ε, κυρίως μάλλον για κρατικές ε, και ακόμη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις μας, μπορείτε, είναι διαθέσιμες, μπορείτε να τις διαβάσετε. Θέλουμε να πούμε πώς ε, είναι σημαντικό αυτό το θέμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το θέμα των κρατικών προμηθειών. Τώρα για να δω μια άλλη παρατήρηση ε, σχετικά με τις διασυνοριακές ε, επενδύσεις και κυρίως τις επενδύσεις που αφορούν σε επιχειρηματικό κεφάλαιο κινδύνου. Ε, επ' αυτού υποβάλαμε μια τροπολογία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσθέτουμε μόνο κάποιες λέξεις, αλλά με την αλλαγή ε, λέμε ότι ε, απελευθερώνονται οι επενδύσει από όποιο κράτος μέλος και αν προέρχονται και ακόμη και αν συνδέονται με κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Η χρηματοπιστωτική αγορά γενικότερα, όχι μόνο η αγορά κεφαλαίου χρηματοπιστωτικού κινδύνου, δείχνουν ότι ε, κάποια μορφή ομοιόμορφοι κανόνε, ενιαίοι κανόνες χρειάζονται κυρίω για τις σοβαρέ μικρομεσαίε επιχειρήσει για να γνωρίζουν ότι υπάρχει περιθώριο αναπτυξιακό, περιθώριο λιγμών και για αυτέ. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους σημεία τα οποία θέλουμε να τονίσουμε, αλλά θα επανέλθουμε σε επόμενη συζήτηση, γιατί ε, καταλαβαίνω και εγώ δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα το απόγευμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί σα ευχαριστούμε κυρία Σφένσον. Ο κύριο Ζουβά είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη για τη δουλειά του. Θα ήθελα όμω να επιμείνω σε μερικές από τις τροπολογίες που κατέθεσα. 52 για την ευρυσιτεχνία. Είναι ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο το οποίο δεν συγκεντρώνει ομοφωνία αλλά φαντάζομαι ότι εδώ θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μια ενισχυμένη συνεργασία. Επιμένω στις τροπολογίες 114, 120, 124 για την πνευματική ιδιοκτησία θεωρώ ότι θα πρέπει να προβάλλουμε, να, θέσουμε, να βάλουμε σε μια καλή θέση αυτό το ζήτημα. Και η τροπολογία 120 πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 222 θα ήθελα κύριε Ισηγητά να λάβετε υπόψη σας την νομιμοφροσύνη και την αμοιβαιότητα στις ε, διεθνείς ανταλλαγές γιατί πολλές φορές ε, επέδειξε αφέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτού του είδους την ε, συνεργασία μιλάει πάντοτε για εταίρους ενώ τελικά πρόκειται για ανταγωνιστές το θέμα λοιπόν της ανταγωνιστικότητας είναι πολύ σημαντικό για τη διασφάλιση του πλούτου μας πριν δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν πρέπει να σας θυμίσω ότι για την Ευρωπαϊκή Ευρεσιτεχνία εμείς στείλαμε ένα σημαντικό μήνυμα κατά την Ολομέλεια του Στρασβούργου όταν ψηφίσαμε την ενισχυμένη συνεργασία. Η κυρία Παμέλα Μπρίντερ που είναι προϊσταμένη στην Γενική Διεύθυνση Β1 της ε, DG Mark της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακαλώ το συντομότερο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο στόχος της Κομισιόν, όπως εξάλλου και ο δικός σας, είναι να έρθουμε εδώ με προτεραιότητες και πρέπει να είναι στοχευμένες, focused για να το πω αγγλικά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε από κοινού τις ε, δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν το συντομότερο από την Κομισιόν και τους συνομοθέτες μέχρι το 2012. Εκτιμάμε ιδιαίτερα τις ε, προσπάθειες ε, των εισηγητών και των τριών εκθέσεων που προσπαθούν να ιεραρχήσουν αυτές τις προτεραιότητες και ο πρόεδρος Μπαρόσο το Φεβρουάριο σε μια διάσκεψη που οργανώσαμε για το Single Market Άκτ εξέφρασε και αυτός ε, την προτίμηση για τις προτεραιότητες. Η δημόσια διαβούλευση και η συζήτηση ολοκληρώνονται σήμερα το βράδυ. Επίσημα είναι η τελευταία μέρα της ε, προθεσμίας διαβούλευσης και η Κομισιόν θα δημοσιεύσει μία έκθεση για το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, αυτών των διαβουλεύσεων ώστε όλοι μας να μπορέσουμε να βασιστούμε στο αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων. Και στα μέσα Απριλίου ελπίζουμε ότι θα εγκρίνουμε την τελική πράξη στην Κομισιόν η οποία μετά θα συνοδεύεται και από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στα τέλη Μαΐου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο και των τριών θεσμικών οργάνων για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποια είναι αυτά τα πρωτεύοντα μέτρα ε, για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Να θυμίσω σύντομα το χρονοδιάγραμμα. Εμείς θα ψηφίσουμε στις 16 Μαρτίου 2011 τον Απρίλιο. Έχουμε αργήσει, αλλά η συζήτηση είναι πολύ ε, σημαντική. Ψηφίζουμε τώρα όλοι. Σας το είχα πει εγώ στην αρχή τη συνεδρίασης. Λοιπόν, μπορεί κανείς να πάει να, να την ψάξει την κάρτα σου. Πω πω την ξέχασε στο Παρίσι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Θα προσθέσουμε λοιπόν μία ψήφο για το ΕΛΚ. Αρχίζουμε με την έκθεση et λοιπόν. Παρακαλώ, ε, μην κάνετε τόσο πολύ θόρυβο. Oh, bah voilà. Donc Δεν είναι κακό μαθήτη τη βρήκε την κάρτα. Εντάξει, μπορείτε και καλύτερα, αλλά ήδη καλά είναι. Λοιπόν, παρακαλώ, όσοι αποχωρούν να μην κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα δώσω το λόγο στην ε, Κριστέν Σαντεμόζε πριν ε, την ε, ψηφοφορία. Πρόκειται για μια πολύ απλή κατάσταση. Έχουμε μόνο δύο τροπολογίες και υποστηρίζω και τις δύο τροπολογίες. Και απαντώ λοιπόν θετικά. Λοιπόν, είναι σύντομη ψηφοφορία. Κανονικά δεν θα ανακύψουν προβλήματα. Θα ψηφίσουμε με ανάταση χειρό, αν συμφωνείτε για το πρώτο θέμα. Παράγραφο 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5α, τροπολογία 2, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Είστε όλοι έτοιμοι? Alors, il manque deux votants. Λείπουν δύο ε, ψηφίσαντε στο. Έχει 14 στο ΕΛΚ. Για ah 30 votants et 30 cartes. 30 κάρτες, 30 ε, ψηφίσαντες, αλλά βλέπουμε 28. Α, εντάξει, λοιπόν, ξανά. Παρακαλώ. Abstention. εγκρίνεται με συντριπτικότατη, με ομοφωνία, όχι συντριπτική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει καμία αποχή, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια, Κρίστελ. Δεύτερη ψηφοφορία τώρα. Alors, deuxième vote. Alors, le vote concernant le rapport de Είναι η ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Καράς. Θα του δώσω το λόγο θα δώσω το λόγο στον κύριο Σουάμπη. δεν χρειάζεται. Ε, απουσιάζει ο κύριος Καράς. Μόλις έμαθα ότι δυστυχώς ε, έπαθε ένα τύχημα σκι πάνω στην πίστα ε, την ώρα που φιλούσε μια Αγγλίδα κυρία. Ε, είναι αληθεύει αυτό. Όχι, ήταν στα αριστερά της. Λοιπόν, ε, αρκετά με τους αστεισμούς. Καλή ανάρρωση του ευχόμαστε και συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Με ανάταση χειρό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, παράγραφο 1, τροπολογία 2. Υπέρ, παρακαλώ. Παράγραφο 1. Παράγραφος, ε, τροπολογία 2 για την παράγραφο 1. Α, θέλετε την κάρτα. Εντάξει, για να είναι όλα σαφέστατα. Λοιπόν, παρακαλώ. Contre. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, πάλι με την ηλεκτρονική σας κάρτα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 3. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 για την παραγραφό 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ας κάνουμε μια επαλήθευση. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν για την τροπολογία, συγγνώμη, 5. Υπέρ κατάλληλη πρόεδρος, αλλά είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Α, όντως, απερίφθη. Μπράβο σας, το είχατε δει ήδη. Ε, τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολ... Παράγραφος 2 τροπολογία 9 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές. τα. Παράγραφος 3, τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 10 παράγραφος 3 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 14. Ζητείτε χωριστή ψηφοφορία. Από το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Για την τροπολογία 14, παράγραφος 3. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15-15 το αποτέλεσμα. Δεύτερο τμήμα. Επίσης θα ψηφίσουμε χωριστά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Α, εντάξει, θα ελέγξουμε. Επανερχόμαστε στην τροπολογία 19 για την παράγραφο 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 ψηφ... την, τροπολογία 19 ψηφίζουμε. Ε, εντάξει, εγκρίνεται, ναι, συγγνώμη. Τροπολογία 20. Διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχει καταπέσει η τροπολογία 24, η 26 έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 8 και τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε. Θα να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 8α τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία Θα έχουμε μία χωριστή ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες. Μα το βλέπετε. Ομοφωνία. Μπράβο, μπράβο στον εισηγητή. Θα πρέπει να τον ε, ενημερώσουμε για να τον εμψυχώσουμε κιόλα. Πάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν. Κύριε Κρόιτσμαν θέλετε να πείτε κάτι. Όχι. Και χάνετε το μικρόφωνο της Προέδρου. Θα είχα μία προφορική τροπολογία για τον συμβιβασμό 1 και θα σας παρουσιάσω αυτή την τροπολογία όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε. Ε, άρα ευθύς αμέσως λέει η Πρόεδρος. Επειδή πρόκειται ε, για μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, σας παρακαλώ να τη διαβάσετε ολόκληρη. Στον Στη συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1 θα ήθελα να προσθέσουμε μία πρόταση ως εξής. Καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μία ειδική πολιτική υπέρ των εποχιακών εργαζομένων. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Πρόκειται για μία προσθήκη στην συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1. Έχετε καμία αντίρρηση προς αυτό? Καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πολιτικές. Ο κύριος Ζουβέν θα μπορούσε να μας διαβάσει ίσως όλη την τροπολογία. Ωραία. Στα αγγλικά καλεί τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν και να προαγάγουν την εκπαίδευση και την, την άσκηση στον τομέα του τουρισμού και των οργανωτών διαστηριοτήτων, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση και εξειδίκευση του ευρωπαϊκού τουρισμού. Επίσης, σε καλή ε, να σημειωθεί η βελτίωση στην αμοιβή αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού, ούτω ώστε ε, να είναι πιο εύκολο και για του εξειδικευμένου εργαζομένου και για όσου ανακυκλώνονται και αλλάζουν σταδιοδρομία να βρούνε δουλειά. Και τώρα αλλάζουμε. Καλεί τα κράτη-μέλη ε, να εκπονήσει μια ειδική πολιτική που θα καλύπτει όλου του εργαζομένου και συνεχίζουμε με το αρχικό κείμενο, υποστηρίζει στεναρά της τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει μια επαγγελματική κάρτα, ένα επαγγελματικό δέλτιο που θα βελτιώσει την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα των ποιοτικών εργαζομένων στον τομέα αυτό και θεωρεί ότι η πρώτη αυτή επαγγελματική κάρτα καλό θα ήταν να εισαχθεί και για τους ε, ξεναγούς ή για τους tour operators μάλλον. Ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Γκέπχαρτ. Äh, Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν την προφορική τροπολογία. Διότι εδώ προσθέτουμε την τελευταία στιγμή κάτι το πάρα πολύ καινούριο και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την, έτσι στα γρήγορα τις επιπτώσεις αυτής της τροπολογίας. Προτείνω να καταθέσετε την τροπολογία αυτή στην Ολομέλεια και επειδή δεν μπορούμε να λάβουμε θέση τώρα, εμείς απορρίπτουμε την προφορική τροπολογία. Ο κύριος Ζιβάν μπορεί να απαντήσει. Κυρία Πρόεδρε και κυρία Γεπχαρτ, ο, η συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1 αποτελεί τον καρπό της ε, συνένωσης πολλών τροπολογιών και εγώ είχα προτείνει μία. και μιλούσαμε για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Δεν είναι ουρανοκατέβατη η πρότασή μου. Βρισκότανε, εμπεριεχόταν σε μία από τις τροπολογίες η οποία χρησιμεύσε για την σύνταξη της ε, συμβιβαστικής τροπολογίας. Μα όπως ε, ήδη το είπα, ε, το να πετάει κανείς κάτι το εντελώς νέο μέσα σε μια συνεδρίαση, κατά τη γνώμη μου είναι λίγο προβληματικό. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους εποχιακούς εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Καλό θα ήταν ο κύριος Ζουβά να παρουσιάσει την πρόταση μέσα στο πλαίσιο της ε, γενικότερης διαδικασίας. Δεν είμαστε κατά, απλώς δεν θέλουμε να δεχθούμε τώρα την προφορική τροπολογία. Ωραία. Πρόκειται για μία last minute προφορική τροπολογία. Θα πρέπει να δούμε πόσες αντιρρήσεις έχουμε. Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω ότι υποστηρίζουμε ως έλκα απόλυτα τον συνάδελφο ε, Ζούβα. Πρόκειται να μπει αυτή, προτείνουμε να μπει αυτή η τροποποίηση μέσα στο γενικότερο πακέτο των τροπολογιών. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Καταλαβαίνω τη θέση της κυρίας Γκέπχαρτ, ε, ε, μα ε, εξεπλάγημεν και εμείς από αυτήν την πρόταση. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τους εποχιακούς εργαζόμενους. Εγώ το βλέπω με καλό μάτι, αλλά αν εσείς το βλέπετε με κακό μάτι, τότε να ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με την Ευελίν. Έτσι όπως διατυπώνεται εδώ είναι ιδιαίτερα αμφίσιμο. Δεν θα έπρεπε εμείς να δημιουργήσουμε διακρίσεις έναντι των εποχιακών εργαζομένων και στο βαθμό που η πρόταση είναι αμφίσιμη και δημιουργεί και πρόβλημα στη μετάφραση ε, θα ήταν καλύτερο να μην το δεχθούμε. Σύμφωνοι. Ε, κοιτάστε κυρία Πρόεδρε, δεν θα τσακωθούμε για το θέμα. Απλώς ήθελα να πω ότι σε ένα θέμα σχετικά με τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για τους εποχιακούς εργαζόμενους διότι πρόκειται για μια οικονομικοκοινωνική πραγματικότητα. Ήθελα λοιπόν να είμαι ρεαλιστής. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση του κυρίου Σβάμπε είναι απόλυτα αποδεκτή. Η κυρία Χούλε Εν αντιθέσει με την κυρία Γκέπχαρτ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να μιλάμε για τους εποχικούς εργαζόμενους γιατί έχουμε προβλήματα σε αυτό το θέμα αλλά αν αυτό μπορεί να μείνει για την Ολομέλεια συμφωνώ ότι θα σας στηρίξουμε. Ε, έχετε το λόγο κύριε Σουάμπ. Με συγχωρείτε γιατί είσαστε πολύ ευγενικοί μαζί μου όσον αφορά την ερμηνεία των κανόνων του Κοινοβουλίου αλλά δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να ε, μπορέσουμε να ε, υποβάλουμε τροπολογία στην Ολομέλεια. Μπορούμε ή δεν μπορούμε. Τα Alors, normalement, on doit pas, quand on regarde le règlement, on ne doit pas déposer d'amendement. Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορούμε να καταθέτουμε τροπολογίες στην τελευταία στιγμή. Μπορούμε να τις ψηφίζουμε εδώ. Και ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θα πρέπει να ψηφιστούν. Ah, oui. Πρέπει ο εισηγητής, ο κύριος Κρόιτσμαν που δεν με ακούει, πρέπει ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής γνωμοδότησης να εκφραστεί. Και να υποστηρίζεται η πρόταση από το 1 δέκατο. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τον συμβιβασμό, μετά την προφορική τροπολογία και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι είναι. Α, δεν είναι και πολύ σαφές εδώ. Voilà. Bon, alors, on va voter θα ψηφίσουμε την συμβιβαστική τροπολογία έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή και μετά θα ψηφίσουμε την τροπολογία του κυρίου Ζουβά και μετά θα δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Σύμφωνοι. Καλή δυο γαϊδά des amendements au rapport Όταν έχουμε έκθεση πρωτοβουλία, είναι σχεδόν αδύνατο να καταθέτει κανείς τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, επιμένω ότι πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες που υπάρχουν στον εσωτερικό κανονισμό και να μην κάνουμε εξαιρέσεις διότι αν ξεκινήσουμε με τις εξαιρέσεις σήμερα ποτέ πια δεν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε τους ισχύοντες κανόνες. Στο βαθμό λοιπόν που έχουμε έστω και μία αντίρρηση δεν λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή την τροπολογία. Έχουμε τουλάχιστον μία ομάδα η οποία έχει αντιρρήσεις με το νέο κανονισμό για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας δεν μπορούμε να καταθέτουμε εμείς προφορικές τροπολογίες την τελευταία στιγμή. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Μα για τον, σύμφωνα με τον κανονισμό είναι αδύνατον κάτι τέτοιο στην Ολομέλεια, αλλά στην Επιτροπή είναι δυνατόν. Αν υπάρχει μια αντίρρηση όμως δεν γίνεται λέει η Πρόεδρος ε, είναι μια ομάδα, απαντάει ο πρόεδρος. Μπορείτε να προτείνετε εσείς ε, στην Επιτροπή Μεταφορών την, ε, την τροπολογία αυτή. μα είναι παράλογο λέει ο κύριος Ζουβά, είναι πολύπλοκος ο κανονισμός λέει η πρόεδρος. Don, ce fort, mais qui est pour la compromis 1 Ποιος είναι υπέρ της τρο... συμβιβαστικής 1. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Και εδώ έχουμε πάλι μία προφορική τροπολογία της τελευταίας στιγμής. Είναι μία τροπολογία της κυρίας Ενάλοβα για την ίδια της ε, την τροπολογία. Ευχαριστώ πρέπει να σας πω ότι δεν θέλω να περιπλέξω την κατάσταση απλούστατα αναφέρομαι στο τελευταίο μέρος της ε, ε, τελικής προτάσεως την οποία προσπαθώ να ε, αποσύρω που λέγει ότι ζητά για αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων ή στην τουριστική βιομηχανία κατά τρόπον ώστε να επιτραπεί εις τους νέους να βρουν δουλειά σε αυτή τη βιομηχανία και να μην υπάρξει μία ε, επιδίνωση των υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται. Αυτό ήτανε. Tomber uniquement ε, la dernière partie de la dernière phrase. Θέλετε μόνο το τελευταίο τμήμα της τελευταίας πρότασης ή όλη την μισή πρόταση. Εάν μου το επιτρέψετε, μόνο το τελευταίο μέρος της τελευταίας φράσης θα εκπέσει, including the provision και από εκεί και πέρα. Δηλαδή και της, ε, την προσφορά του δυνατοτήτων ε, Παροχή υπηρεσιών για τις τουριστικές υπηρεσίες από τρίτε χώρε. Αντιρρήσει επ' αυτού. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Δεν το μπορώ να το δεχτώ και ζητώ να απορριφθεί. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 έτσι όπως διατυπώθηκε πριν από την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Καθ' ολοκληρία ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 του κυρίου Ζουβά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 για την παράγραφο 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται διορθώνει την πρόεδρος. Παράγραφος 1 γ. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19, παράγραφος 1 δέλτα σε πολλά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Κύριε Σβάμπ, εσείς είστε μεταξύ δύο θέσεων. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβιβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές για να το επαληθεύσουμε ψηφίζουμε κατά περίπτωση λοιπόν αρχίζει η πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται παράγραφος 3 συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3β τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά α, να το επαληθεύσουμε πέρα στις α, επαληθεύουμε την 35 πέρα της ψηφοφορίες Απορρίπτεται. 40. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 και 42. Υπέρ. Κατά. Έχει καταπέσει, έχει καταπέσει. Συγγνώμη, δεν πρόσεξα, λέει η Πρόεδρο. Τροπολογία 43. Και αυτή έχει καταπέσει. 44. Προσθήκη. Υπέρ τη 44. Κατά. Αποχές. Νομίζω να, ότι εγκρίθηκε. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 48. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά και εδώ να το επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 45 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 49. πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4β. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. 4β λοιπόν, τροπολογία 53, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 56, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 57 ψηφίζουμε σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά 57 Πρώτο τμήμα. Εγώ έχω δύο. Ναι, ναι, δύο τμήματα υπάρχουν. Βεβαίω, πρόκειται για χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 57. Α, εδώ μου λένε ότι είναι κακοφτιαγμένος ο κατάλογος ψηφοφορίας. μάλιστα ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα και φτάνει τότε. Τώρα η τροπολογία είναι του κυρίου Εκ. Ο κατάλογος ψηφοφορίες δεν ήταν σωστό Ψηφίσαμε συνολικά λοιπόν τον 57. Μα εγώ έχω μία λίστα με χωριστή ψηφοφορία κυρία Πρόεδρε. εδώ είμαστε πολύ μπερδεμένοι με την ψηφοφορία σήμερα. Μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Ψηφίσαμε το πρώτο τμήμα, άρα ψηφίζουμε το δεύτερο. Για τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς. Ναι, ναι, ναι, λέει η πρόεδρος, το πρώτο τμήμα το ψηφίσαμε και θα ψηφίσουμε το δεύτερο, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Πέρασε λοιπόν το πρώτο τμήμα και απορρίπτεται το δεύτερο. Θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Παράγραφος 4 γάμα 58 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, 60 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρες ψηφοφορίες.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 Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρασε ψηφοφορίες και εγκρίνεται. Μπράβο. Τελευταία ψηφοφορία. Έκθεση της κυρίας Ανάλογα. Τροπολογία 1 για το παράγραφο 1 υπέρ. 1, Και πάλι υπάρχουν λάθη στον κατάλογο ψηφοφορίας εδώ. Σε δύο τμήματα η ψηφοφορία λέει εδώ. Στην παράγραφο 1 είμαστε πάντως, ε, συμβαστική, ένα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα τώρα, με την προσθήκη της λέξης constantly. Παρακαλώ. Κατά. Ίσως πρέπει να κάνουμε την επαλήθευση, δεν είμαι σίγουρη. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της πρώτης συμβαστική. Με την κάρτα, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Ωραία. Παράγραφος 2 τώρα. Ένα τμήμα. Υπάρχει μία ή, ή τρεις προφορικές τροπολογίες, γιατί γράφει τρεις εδώ. υπήρχε από το Λουί Γκρέκ μια προφορική τροπολογία, αλλά υπάρχει μέσα στον κατάλογο, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ψηφίζουμε για τη δεύτερη παράγραφο, νέα, με τις τρεις ε, τροπολογίες ε, που έχουν ήδη καταγραφεί. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 4. Τροπολογία 4, έτσι υπέρ κατά επαλήθευση νομίζω χρειαζόμαστε άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν πέρας τώρα Et rejeté. Απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 2 γάμα τώρα, υπέρ. Είναι η τροπολογία 5. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Alors, Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πάμε στην ε, τρίτη παράγραφο τροπολογία 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η τροπολογία 9 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 3 γ, τροπολογία. Έχουμε κατά τμήματα μάλλον ψηφοφορία και για αυτή την παράγραφο. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 4, συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην παράγραφο 5, συμβαστική υπαριθμό 4, υπέρ. Ah, Alors, speed vote. Πάλι είναι κατά τμήματα η ψηφοφορία, διορθώνει η πρόεδρος το πρώτο κομμάτι, ακέραιο το κείμενο, χωρίς το of the social and economic impacts. Υπέρ, για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Κατά. Μάλιστα. Α κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για να είναι σαφέστερα τα πράγματα. Θα ψηφίσουμε για τη συμβαστική. τέσσερα, πέμπτη παράγραφος, δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Le vote est clos. Et c'est rejeté. Απορρίπτεται. Et nous ε, τώρα πάμε στο 17. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ε, η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Να κάνουμε παλήθευση. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την παράγραφο 5β. 5Γ μάλλον, η τροπολογία 19. Πέραση τη ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Κατόπιν, ε, παράγραφος 6. Είναι ε, ομού η τροπολογία 20 και 21. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 7, συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7α, ε, η τροπολογία 23 με μια προφορική τροπολογία που έχει κατατεθεί και καταχωρηθεί υπέρ, κατά, άποχες. Ε, δεν σηκώνετε καλά το χέρι, δεν σας βλέπω ξανά υπέρ, κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η επόμενη και πάμε στην 24 παρακαλώ, παράγραφος 7, 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέλος. Θα ε, προβούμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. της νομοδότησης ε, ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητηρία. Κυρία Σεχνάλοβα. Τελειώσαμε και τις ψηφοφορίες. Η πρόεδρο ζητά συγγνώμη. Ε, είχαμε ε, κάποιες δυσκολίες με τον κατάλογο ψηφοφορίας, δεν είχαμε το σωστό κατάλογο. Τέλος πάντων θα εκχωρήσω τώρα την Προεδρία στη συνάδελφό μου. half an hour late. We're, half an hour late at the moment. Merci. Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour late at the moment, so we will start immediately and I want to... Ε, συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε ευθύς αμέσως. Ο κύριος Βιμ Βαντεγκάμπο, εισηγητής μας, θα πάρει το λόγο, ούτως ώστε να μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας για τον έλεγχο της αγοράς για τα δίκυκλα και τρίκυκλα ε, οχήματα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα κτλ. Παρακαλώ να είστε σύντομος, ακριβείς, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. So please, Mr. Van Dekker. Uh, mevrouw de voorzitter. Κύριε Φαντεκάμπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, καλό απόγευμα σε όλους. Χαίρομαι για την προσέλευση. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι σήμερα. Ε, κυρία Πρόεδρε, το έγγραφο εργασίας μας ε, νομίζω δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσει. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξη και τη βοήθεια τους. Ε, τις ε, προσεχείς εβδομάδες και μήνες θα κληθούμε να λάβουμε διάφορες αποφάσεις προς το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. πρέπει να ε, αποφασίσουμε επίσης ε, για τα κριτήρια, τα περιβαλλοντικά κριτήρια και κυρίως ε, για τις προθεσμίες θέσεις ισχύω των προτύπων 5 και 6, ευρώ 5 και 6. Επίσης να αποφασίσουμε για τα συστήματα πέδησης. Είναι λίγαν τεχνικό το ζήτημα. Ε, θα πρέπει εν συντομία να αποφασίσουμε πότε θα ε, ε, γίνουν υποχρεωτικά αυτά τα νέα συστήματα παίδησης. Επίσης θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σχετικά με τα διαγνωστικά συστήματα του οχήματος και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα λειτουργίας του οχήματος. Επίσης, θα πρέπει να για τους ε, ε, εξισοδοτημένους ε, αντιπροσώπους να αρχίσουν να ισχύουν οι νέες διατάξεις για τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων κατόπιν να αποφασίσουμε το συνολικό τροχνοδιάγραμμα πότε θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τα επιμέρους μέτρα κατόπιν θα εξετάσουμε αν μπορούμε να απλουστεύσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα επίσης Πρόεδρε να αναφέρω ότι στις, συναντηθήκαμε στις 28 Ιανουαρίου συναντηθήκαμε στις κάτω χώρες για να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυ τα συστήματα αντιεμπλοκή κατά την πέδηση, τα λεγόμενα ABS, και την περασμένη εβδομάδα ε, μεταβήκαμε στην Μπολόνια και την Ε, και επισκεφτήκαμε πολλά εργοστάσια Κατόπιν, απευθυνόμενο ε, στου ε, σκιώδει εισηγητέ, θα ήθελα να σα πω ότι η Επιτροπή Μεταφορών ε, και Τουρισμού έχει ήδη εγκρίνει την γνωμοδότησή τη. εκεί περιέχονται ε, πολυάριθμε, πολύτιμε παρατηρήσει για το σχέδιο κανονισμού. Σε αυτή την ίδια γνωμοδότηση προβλέπονται επίση διάφορα κριτήρια που θέλει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα οχήματα, κριτήρια αυστηρότερα σε σχέση ε, με τις αρχικές προθέσεις. Ιδού και κλείνω. Ε, δεν έχω άλλα εισαγωγικά σχόλια. Thank you very much. And the next... Ευχαριστώ. Ο, η, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Αλλά βλέπω ότι έχει φύγει. Άρα θα επανακάμψει. Ο κύριος Μάντερς επίσης δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρούλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ δεν είναι μόνο ευγένεια διότι είναι κάτι που με ενδιαφέρει πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο θέμα που θέτει όλα τα καυτά ερωτήματα και ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και εγώ ασχολούμαι ιδίως με ε, το scope διότι ξέρετε ότι ε, δεν γνωρίζω αρκετά τον όρο e-bikes, δηλαδή ε, μοτοποδήλατα τα οποία έχουν και κινητήρα και πεντάλια. Είναι κάτι νέο και πολύ ε, προχωρημένο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται και δεν πρέπει να υπερφορτώσουμε με γραφή αυτό το συγκεκριμένο θέμα αλλά σύμφωνο ότι περιβαντολοντολογικά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα ισχύσει και να δούμε και το χρονοδιάγραμμα δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε το χρονοδιάγραμμα για να μην υπάρχουν διάφορα χρονοδιαγράμματα τα οποία συγκρούονται. Με, δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω στις επισκέψεις θα υπάρξει και μία το Μάιο όπου δεν θα μπορέσω να παραστώ αλλά σε όλες τις εκδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται στο Κοινοβούλιο συμμετέχω και ο τομέας αυτός με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως έχω κάνει και ορισμένες συζητήσεις και πιστεύω ότι σύντομα θα συμφωνήσουμε σε μία ενιαία θέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον συνάδελφο για τη θαυμάσια επίσκεψη που οργανώθηκε στην Ιταλία και πραγματικά μάθαμε πολλά. Θέλω να προσθέσω κάτι Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του, αλλά αν είναι δυνατόν θέλω να δω εάν μπορούμε να προτείνουμε και την προέλευση, διότι όπως άκουσα υπάρχουν πολλές, πολλά παραποιημένα μοτοποδήλατα τα οποία εισάγονται από πολλά μέλη του κόσμου και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οδηγούμε μια πραγματική βέσπα και όχι κάτι κινέζικο. Ε, μετά η κυρία Τέ που αντικαθιστά το Μάλκορ Χάμπον. Έχω μεταμορφωθεί σε Μάλκομ Χάρμπερ. Υποστηρίζει τον κύριο Φαντεν Κάμπ και τις προτάσεις του εγγράφου του επειδή υπάρχουν ε, διάφορε ημερομηνίε εφαρμογή για τι επιμέρου απαιτήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται αναθεώρηση τη εφαρμογή ε, ε, και προτιμούμε να αναθεωρηθεί και να απλουστευθεί το χρονοδιάγραμμα. Θα είναι έτσι απλούστερα τα πράγματα για όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Ο κύριο Χάρμπορ θεωρεί ότι οι μακροπρόθεσμε απαιτήσει θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εξολόγηση αντικτύπου. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητείται να δώσει εξηγήσει για το θέμα των τεχνικών πληροφοριών και του χειρισμού, τη διαχείριση των τεχνικών τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτούς που επιδιορθώνουν τα ε, οχήματα αυτά και επίσης ε, ε, ζητώ συγγνώμη γιατί διαβάζω τις σημειώσεις κάποιου άλλου και δεν είμαι σίγουρη ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση έχει κάνει προτάσει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και ελπίζει ο κύριο Χάρμπουρο ότι θα ισχύσουν ενιαίε διατόξει για όλα τα δίκυκλα οχήματα. Ε, κοιτάξτε, λέει η πρόεδρο, είναι η τυχερή σα ημέρα και η τυχερή του κυρίου Χάρμπορ. Ποτέ δεν ήταν τόσο όμορφο ο κύριο Χάρμπορ όπω είσαστε εσεί. Ε, κυρία Ευχαριστώ και εγώ με, τα, μετουσιώνομαι γιατί ο συνάδελφος Βέστφαλ ε, βρίσκεται σε μία άλλη επιτροπή ε, για ψηφοφορίες και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω. Μου έδωσε και ένα γραπτό κείμενο γι' αυτό και είναι πιο απλό να το παρουσιάσω ευχαριστεί για, την, ε, για αυτό το ενδιαφέρον για το φάκελο και ε, συμμετείχε σε, όλες, ε, σε όλα τα θέματα. Είναι κάτι το οποίο θεωρεί πολύ ικανοποιητικό και όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας θεωρεί ότι είναι καλό ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στο κείμενο διότι τα θεωρεί πολύ σημαντικά και τώρα θα σας διαβάσω το σημείωμα της συναδέλφου δηλαδή ότι όποιος ε, θέλει να κινείται στο μέλλον με δίκυκλο και όχι με αυτοκίνητο αποδεικνύεται πολύ ε, πιο θετικό με την αύξηση των δικύκλων ιδίως η στις ε, τις αστικές περιοχές όπου υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Θα έπρεπε καταρχήν να μου ε, επιτρέψετε να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και εδώ στηρίζω την, ε, τα κίνητρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα 15-20 χρόνια πρέπει να μπορέσει να ισχύσει αυτή η νομοθεσία για να αισθάνονται ασφάλεια και οι κατασκευαστές και ε, αυτά, ε, αυτός ο κλάδος καλύπτεται περισσότερο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, υπάρχουν ίσως λίγες ε, ε, επιχειρήσεις αλλά δεν πρόκειται για μία αμυγός ευρωπαϊκή αγορά αλλά για μία ενιαία αγορά και γι' αυτό οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις είναι απαραίτητες και πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του κανονισμού ε, θα έχουν επιπτώσεις σε ένα τομέα ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είχε φυγεί και επιπλέον των προηγουμένων σημείων θεωρώ ότι και αν είναι ισοσκελισμένος ε, ε, ο ε, ισοσκελμένη οδηγία η κίνηση θα είναι μονοπλευρή και αυτό νομίζω ότι εκφράζεται πολύ επίοικος διότι πιστεύω ότι πολλές προσπάθειες θα αποτύχουν και πρέπει να δούμε αν πρέπει να το επιτρέψουμε διότι ότι αυτά τα οχήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες της εποχές, εποχής, να είναι ε, πιο ασφαλή και ε, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και αυτές είναι οι επιταγές που οι καταναλωτές μας απευθύνουν ε, και όλα αυτά θα πρέπει να επιτρέψουν στην βιομηχανία να είναι και οικονομικό θετική και φιλική προς το περιβάλλον. Ορισμένες λοιπόν κατηγορίες πρέπει να είναι πιο σαφείς τόσο ε, για τα ε, ελαφρώς ε, μηχανοκίνητα οχήματα όσο και για τις εξαιρέσει από τον κανονισμό διότι το ερώτημα είναι αν πρέπει να υπάρξουν ειδικέ διατάξεις για ορισμένα προϊόντα ή αν υπάρχει τρόπος να τα οριοθετήσουμε με κάποιο τρόπο. Και εδώ ανεφάρουμε στο ITV ή ε, e-bikes ε, και πρέπει να σας πω δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί τύποι οχημάτων διότι εγώ δεν τους προτιμώ. Επίσης ε, πρέπει να γνωρίζουμε πέραν του ποσοστού του της αγοράς που χρησιμοποιούνται τα οχήματα αυτά και η κατηγορία λάμδα δεν συναντάται τόσο πολύ στο δικό σύστημα όσο άλλα οχήματα παρόλα αυτά έχει πολύ υψηλές εκπομπές και οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Άρα θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια βελτίωση ε, παρόλο που ήδη έχουν γίνει αρκετά και έχω ακούσει από πολλούς ότι ε, τεχνικά ορισμένα από αυτά τα οχήματα είναι πεπαλαιωμένα όσον αφορά ε, τον φιλικό υλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα και επίσης και όσον αφορά το σύστημα παιδίσεως. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε πόσοι είναι οι νεκροί από, τις, ε, ε, από αυτοκινητιστικά και πρέπει να δούμε ότι ο αριθμός των νεκρών από ατυχήματα με δίκυκλα, με εμπλοκή δικύκλου αποδεικνύει ότι χρειάζεται μία βελτίωση του συστήματος διότι μπορεί να έχουμε προβλέψει το ABS για τα αυτοκίνητα και να θεωρούμε ότι αυτό λύνει το πρόβλημά μας αλλά δεν ισχύει διότι ε, όταν υπάρξει χρήση του συστήματος ABS στα μοτοποδήλατα θα μπορέσουν επίσης επίσης να περιοριστούν τα θανατηφόρα ατυχήματα ένα μοτοποδήλατο δεν είναι αυτοκίνητο δεν μπορώ να ανοίξω τη μηχανή και να περιλάβω όλες τις τεχνικές προόδους στα δίκυκλα χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και λεπτότητα αλλά υπάρχουν δυνατότητες βελτιώσεως και θα πρέπει να μπορέσει κανείς να αλλάξει και την δομή και την τιμή του οχήματος για να μπορέσει να δεχθεί τις τεχνικές αλλαγές διότι διαφορετικά σε, δύο, σε μερικά χρόνια δεν θα μοιάζει καθόλου με τη, στη σημερινή του μορφή. Εμείς όμως εδώ ζητάμε να υπάρξει μία ισχύς των διατάξεων για 15-20 χρόνια και αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ασφαλείας. Πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ως πιο χρήσιμο καθοριστικό στοιχείο την ασφάλεια και να προβούμε σε μία βελτίωση της ασφαλείας των οχημάτων αυτών για να μειώσουμε τον αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων διότι διαφορετικά ε, αν αυτό δεν επιτευχθεί θα μπορέσει να συνεπιφέρει και οι οικονομικές ζημίες και παρόλο που το απέφχομαι ε, θέλω να συνεργαστώ αγαπητοί ε, συνεργάτες μαζί σας για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Είμαι όμως πολύ επιφυλακτικός και θέλω να πω στον κύριο Κάρφο ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε συνένεση. Σας ευχαριστώ όμως για το έγγραφο εργασίας σας και για το πνεύμα συνεργασίας σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκέπχαρντ. Ο κύριος Μαρτίνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει τώρα τον λόγο. Thank you and Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσουμε το θέμα αυτό. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες ε, του εισηγητή και των ε, σχεδόν εισηγητών, γιατί κατάφεραν να εξοικειωθούν με ένα με μια τόσο περίπλοκη και τεχνική πρόταση. Προφανώς ε, ε, καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασίας είμαστε στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες για την αρχική μας πρόταση. Χαίρομαι πάντως διότι με το έγγραφο εργασίας που συζητείτε σήμερα θα, θα εστιάσετε την προσοχή σας στα βασικότερα ε, σημεία προ απόφαση. Πρόεδρος, ε, είμαστε πάρα πολύ έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά θα δώσω τη δυνατότητα στην κυρία Γιάκομπ, αν θέλει, να παρέμβει για λίγα λεπτά. Θέλετε? Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, ευχαριστώ και τον κύριο Βάντερ Κάμπ για την έκθεση. Η εργασίες της ομάδας εργασίας συνεχίζονται. Έχουμε δύο σχέδια που εκκρεμούν προς έγκριση. Ένα για τα τρακτέρ και ένα για την κατηγορία ε προσπαθούμε να διαχειριστούμε αντίστοιχα τους κανόνες, τους ε, κανόνες των δύο κατηγοριών που μοιάζουν μεταξύ τους. Η Προεδρία θα αποφασιστούν τα μέτρα αυτά και να το λάβετε υπόψη σας όταν θα πρέπει να αποφασίσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντερκάμπ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκεώδεις εισηγητές όπως επίσης και το Συμβούλιο και την Κομισιόν για τις παρατηρήσεις τους. Θα συνεχίσω την εξέταση αυτού του τεχνικού πραγματικά θέματος Αν βέβαια ε, η κυρία, που αντικαθιστά τον ε, κύριο Χάρμπορντ συνεχίσει να τον αντικαθιστά, εγώ θα είμαι πανευτυχής. Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα υπάρχουν πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα. Υπάρχουν όμως ε, βιομηχανίες που θέλουν συνολικά μία έγκριση για την ευρωπαϊκή αγορά. Με την κυρία Ρούλε και τον κύριο Χάρμπουργκ θα πρέπει να το σκεφτούμε για να δούμε ποια θα είναι η μοίρα των ηλεκτρικών ποδηλάτων διότι η απόφαση αυτή θα έχει πολλές επιπτώσεις για το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό γιατί συνδέεται με τα γενικότερα μέτρα για το περιβάλλον. Για την ονομασία προέλευσης. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό έχει τη θέση του σε αυτό το κείμενο. Πρέπει να το συζητήσουμε με την Επιτροπή για να δούμε αν μπορούμε να προσθέσουμε και αυτή τη διάσταση ή όχι. Σίγουρα υπάρχουν ένα σωρό ψεύτικα, ε, ε, ένα σωρό σκούτερ μαϊμούδες ε, ε, των Ιταλικών ε, στην αγορά και πρέπει να το περιορίσουμε. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρ για την τόσο τεχνική σας παρέμβαση και η παρατήρηση της κυρίας Βέσφαλτ θα, είναι, θα ληφθεί υπόψη αυτούσια. Για το θέμα των αυτοκινητιστικών ε, δυστυχημάτων και τους κανόνες φρεναρίσματος και αυτά θα ληφθούν υπόψη. Θα πάμε στην Έση και στο Στρασβούργο για αντίστοιχε επισκέψεις και θα έχετε τις λεπτομέρειες αυτών των δύο επισκέψεων το συντομότερο. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο την Επιτροπή. Στην Πολόνια, στο εργοστάσιο της Δουκάτη, μας μίλησαν για μια νέα αντίληψη που ονομάζεται traction control και που δεν την έχουμε στην πρόταση για τις προδιαγραφές και για την παραλαβή. Μπορεί να μας απαντήσει η Κομισιόν τι κάνουμε με αυτό το tract control. Θα παρουσιάσουμε στα τέλη Μαρτίου, αφού ακούσουμε όλη την Επιτροπή, την τελική έκθεση. Θέλουμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο σύντομα, οπότε ίσως να διμερώς να το συζητούσατε. Το επόμενο σημείο είναι η πολιτική ραδιοφάσματος. Κανονικά θα έπρεπε την περασμένη φορά να το έχουμε συζητήσει, να το έχουμε ολοκληρώσει το θέμα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορχόλα την συγγήτρια. Το πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος λοιπόν ο στόχος είναι η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό αυτό βήμα ούτως ώστε να έχουμε τη βέλτιστη οικονομική ε, και κοινωνική χρήση αυτού του δημοσίου αγαθού και η πολιτική ραδιοφάσματος ε, είναι στο κέντρο του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμβληματικής αυτής της πρωτοβουλίας και σχετίζεται και με πολλούς άλλους στόχους πολιτικής στα πλαίσια του θεματολογίου 2020. Ε, δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μια συντονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να τονώσει την οικονομία έως και 44 δις ευρώ. Ε, η αποτελεσματική κατανομή και διαχείριση του ραδιοφάσματος προσφέρει ε, κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά στους Ευρωπαίους πολίτες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας ε, επίσης ε, συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας εύρωστης ενία αγοράς για αγαθά και για υπηρεσίες. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η κινητή τη τηλεφωνία τα τελευταία τρία χρόνια ε, είχε κατακόρυφη αύξηση και συνεχίζεται αυτή η τάση σήμερα. Τα τέιμπλετς, οι φορητοί υπολογιστές κυκλοφορούν όλο ένα και περισσότερο στην αγορά με αντίστοιχες ταχύτητες. Επίσης, βασικό κομμάτι καινοτομίας είναι ναι, οι ευρωζενικές συνδέσεις για τις διοικητικές υπηρεσίες, για την τηλεϊατρική κτλ. Έτσι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους αποτελεσματικές καινοτόμες νέες τεχνολογίες. Δεν μπορούμε να είμαστε ουραγοί. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερο ραδιοφάσμα για, την ε, για το ευρυζωνικό κινητό δίκτυο. Επίσης, η ανάπτυξη νέων δικτύων και νέων συσκευών για τους καταναλωτές θα μειωθεί με την ανακατανομή του φάσματος, θα μειωθούν οι διασυνοριακές παρεμβολές, θα ενισχυθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα τονωθεί και η έρευνα και η καινοτομία. Θα ήθελα να σας πω πως συμφωνώ ε, με τον κύριο Χιόκμαρ, τον εισηγητή της ε, καθήλυνα αρμόδιας επιτροπής, ε, δηλαδή ισχυρίζεται ότι πρέπει να έχουμε ε, φιλόδοξους στόχους ένα αλλά να μην αποτελεί αυτό ακρογωνίο λάθος της πολιτικής ραδιοφάσματος. πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Παραδείγματος χάρη τη ΣΥΠΑ, ε, που είναι ανταγωνιστές Ευρωπαϊκής Ένωση έχει κατανεμηθεί μεγάλο κομμάτι του ραδιοφάσματος για τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας. Ο στόχο είναι να ε, ε, δοθούν για τις κινητές, τις ασύρματες υπηρεσίες τουλάχιστον 1200 MHz. Κατόπιν ε, ε, από τα 790 MHz μέχρι τα 862 MHz αυτή είναι μια ζώνη βασική σημασία για να υλοποιηθεί το ψηφιακό θεματολόγιο της Ένωσης. Η διαδικασία πρέπει να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν, αμελητή και σίγουρα όχι αργότερα μετά δηλαδή το 2013. Ε, το στρατηγικό έγγραφο του προγράμματος πολιτικής ραδιοφάσματος επιζητά ε, ε, μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Για ε, το 2014 και μετά οι βιομηχανίες ζητούν ρυθμιστική ασφάλεια και για όσοι επιχειρήσεις βασίζονται στη χρήση του ραδιοφάσματος είναι ευνοητό ότι καλό θα ήταν να ε, ε, γνωρίζουν τι θα συμβεί μετά το 2015 γιατί χρειάζονται ε, υψηλέ επενδύσεις στη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος και αυτό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση άρα θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα ισχύει μετά το 2015. Για τι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπέ τώρα στην Επιτροπή Πολιτισμού ακούστηκε μια αντίεπιχειρήση επιχειρηματολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν θέσει επιβλαβής σε επιπτώσει, στι οποίε αναφέρθηκε αυτή η Επιτροπή. Το αντίθετο, ε, θα έχουμε περισσότερα πολιτιστικά αγαθά χρησιμοποιώντα νέε τεχνολογίε και η τηλεόραση θα υπάρχει σε όλε τι πλατφόρμες, τεχνολογικέ πλατφόρμε, ακόμη και στην κινητή. Επίση, ε, για τι ασύρματε ευρυζωνικέ συνδέσει, χρειάζεται περισσότερο ε, ραδιοφάσμα, διότι έχουμε εκατοντάδε κανάλια ήδη, αναπτύσσονται νέε τεχνολογίε σε διαρκώ και είναι πιο αποτελεσματική η αναμετάδοση. Αυτή είναι η τροπολογία 60. Ε, στο μέλλον ε, ε, θα μπορέσουν για τις εκπομπές να περάσουν όλοι στη χρήση της ζώνης μέχρι τα 2 GHz και να μειωθεί αν γίνεται ε, να διευρυνθεί η χρήση της ζώνης μέχρι τα 300 ε, MHz και έχουμε και την, ε, στο 2016 την παγκόσμια διάσκεψη για αυτό το θέμα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τι προτάσει που θα κατεβάσουμε για να δούμε και τι θα γίνει μετά το 2020. Επίση, τροπολογία 16, αντισταθμιστικά μέτρα. Ε, για τα για τις ασύρματες συνδέσεις. Ε, όλοι αποσκοπούν σε ένα εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, ούτω ώστε τα ασύρματα μικρόφωνα μπορέσουν να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ε, στις ίδιες συχνότητες όμως ανά την Ευρώπη. Προτείνω να προωθήσουμε και εμείς την εναρμονισμένη αυτή η ζώνη υψηλών συχνοτήτων ε, άνω του 1 GHz. Αυτή είναι η τροπολογία 18. Ε, κατόπιν, ε, μάλλον τώρα ε, οι συχνότητες διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο και από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα για τους καλλιτέχνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν, ο ανταγωνισμός εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την σημασία του ανταγωνισμού, τόσο ώστε να είναι καλές οι τιμές για τους καταναλωτές και ε, να ευνοείται η καινοτομία. Ε, τώρα, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο φάσμα των 800 MHz, δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Για το 2020 και σε ευρυζωνικές ε, συνδέσεις. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε ε, τις προτάσεις, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι διαφέρει η κατάσταση από το ένα κράτος στο άλλο. Γι' αυτό και προτείνω να, το, να επαφείται αυτό στη διακριτική ευχέρεια του κράτους. Δηλαδή, για τις δημοπρασίες τη ζώνη των 800 MHz θα πρέπει να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη και καθώς και για τους επιμέρους ειδικού στόχους. Αυτή είναι η τροπολογία 17. Ε, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα πολιτικής ε, ραδιοφάσματος ε, στην τροπολογία 11 και 7 ε, θα πρέπει να καλύπτει και τους παρόχους της κινητής τηλεφωνίας και το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει το ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι οι όροι ανταγωνισμού. Κάποιοι ε, φορείς ε, αναφέρθηκαν ε, στις παρεμβολές. Δεν είμαι σίγουρη ότι ένα στρατηγικό έγγραφο είναι το κατα... ο κατάλληλος χώρος για να μιλήσουμε για τις παρεμβολές, για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα πρότυπα για να καταπολεμηθούν οι παρεμβολές. Η ίδια η εναρμόνιση ούτως ή άλλως ε, θα λύσει αυτό το πρόβλημα των παρεμβολών στις ε, μεθοριακές περιοχές. Όταν ε, καθαρίζουμε μια ζώνη συχνοτήτων είναι προφανές ότι θα ανακύψουν προβλήματα και κόστος για τη βιομηχανία. Πρέπει να προσαρμοστούν σε άλλες ζώνες. Τα κράτη-μέλη θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για να αντισταθμίσουν τις προσπάθειες, το βάρος αν θέλετε που θα φέρουν οι φορείς της βιομηχανίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξαιρετική έκθεση. Εγώ συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό τις ε, θέσεις σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρεμβαίνει κανείς ε, στο ραδιοφάσμα και θα πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό στρατηγικό πρόγραμμα σχετικά. Συμφωνούμε σε αυτό. Πιστεύω όμως ότι είναι εξίσου σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι συχνότητες, οι ραδιοφωνικές συχνότητες είναι μία, ένας κριτικός πόρος. Οι θέσεις μας πρέπει να είναι σαφείς και τα αιτήματά μας εξίσου. Και η ομάδα μου συμφωνεί σε αυτό. Θα πρέπει το πρόγραμμα να εγγυάται την δυνατότητα των επιχειρήσεων και αυτών που παρέχουν πληροφορίες υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα ενδιαφέροντα της κοινής, ε, τα συμφέροντα της κοινής γνώμης και των καταναλωτών. Για παράδειγμα, τα δημόσια ΜΜΕ βρίσκονται σε μια λεπτή κατάσταση και αυτό μας το παρουσίασε η σχετική γνώμη της Ήτρε. Πρέπει να έχουμε καθαρά υπόψη μας όταν αποφασίζουμε για τέτοια πράγματα και την κατοχήρωση των δημοσίων υπηρεσιών, στην προκειμένη περίπτωση των εθνικών τηλεοπτικών δικτύων. Θα πρέπει θα, πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται στα κράτη-μέλη αλλά οι διαφορές είναι τεράστιες όσον αφορά στα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα και πόσο μάλλον δηλαδή των δημοσίων υπηρεσιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω διότι για μένα υπάρχουν δύο θέματα σε αυτήν την ε, οδηγία. Καταρχήν το θέμα των ε, συχνοτήτων και ε, η κατανομή τους διότι αντιλαμβάνομαι ότι οι δέσμοι των 300 με έχει προβλεφθεί να ανοιχθεί στον ανταγωνισμό βαθμιαίος το 2015 για να μπορέσουν όλοι να προχωρήσουν και να μπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο ε, να υπάρξουν ε, συνδέσεις και να υπάρξει ένα διαδίκτυο σε αυτές τις συχνώσεις γιατί σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι τελείως παραγωγικό, αντιπαραγωγικό και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ε, ευρυζώνια δέσμη για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αφού όμως εξασφαλίσουμε ότι από πλευράς κόστος και κόστους και τεχνικών προδιαγραφών δεν θα είναι εις βάρος των τηλεοπτικών εκπομπών που ενδιαφέρουν το 60% του πληθυσμού. Τα υπόλοιπα βέβαια μπορούν όλο και να βελτιωθούν αλλά μακροπρόθεσμα δεν πρέπει να προτιμήσουμε ορισμένες τεχνολογίες αλλά να κοιτάξουμε ποιο σύστημα θα είναι πιο αποτελεσματικό. Θα μπορούσαν βέβαια να προταθούν και άλλες ε, συχνότητες ε, για την τηλεόραση και για άλλες εκπομπές που τώρα αντικρούονται. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια όπως είπε η κυρία Μόζε. Δηλαδή ε, πρέπει να δούμε ποια είναι οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Διότι παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, στο Βερολίνο, τα μεγάλα αστικά κέντρα χρειάζονται μια καλή δυνατότητα διάδοση του συστήματος και με το ευρυζωνικό σύστημα αυτό επιτρέπεται. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις διαφορές μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων διότι για, τις για την μεσαία τάξη πρέπει να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις ε, για την χρήση του ευρυζωνικού συστήματος. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ε, είναι υποχρεωμένες πρώτα να δημιουργήσουν δυνατότητες ε, διαδικτυακές ή στην Ήπεθρο και μετά να προχωρήσουν στις πόλους. Στην Γερμανία ίσως το σύστημα είναι διαφορετικό, αλλά δεν είναι προφανές ότι σε όλες τις χώρες ε, της Ευρώπης υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν ε, ε, δεν υπάρχει μία κρατική χρηματοδότηση πρέπει να δούμε αν και εκεί μπορεί κανείς να προχωρήσει σε έναν εμπλουτισμό της υπαίθρου ώστε να μπορέσει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Επίσης ε, θα χρειαστεί μεγαλύτερη εναρμόνιση και καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την κατάρτιση τεχνικών παραμέτρων για να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών ε, ότι πρέπει να υπάρξει μία διασύνδεση χωρίς παρεμβολές μεταξύ ε, πηγείων σταθερών σταθμών και κινητών των υπηρεσιών. Επίσης πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των συχνοτήτων εκπομπών κατά τρόπον όλα τα ιατρικά μηχανήματα να βασίζονται στις ίδιες προδιαγραφές σε όλη την Ευρώπη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών και να ε, αυξηθεί και η δυνατότητα επιλογής ε, των πολιτών. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες. Λογικό ακούγεται να εναρμονίσουμε τη χρήση του ραδιοφάσματος στο μέτρο του δυνατού στην Ευρώπη, ώστε οι κατασκευαστές ε, να μπορούν να ε, φτιάχνουν συσκευές για ε, πολλά εκατομμύρια καταναλωτών. Ε, ε, επίσης συμφωνώ με την κυρία Σάλτεμος. Ε, όταν θέλουμε να θεσπίσουμε τεχνικούς κανόνες για την κάλυψη, για το, γενικότερα για το ραδιοφάσμα, νομίζω ότι πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και να επευθύνει τη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους. Είναι προφανές ότι ισχύουν άλλοι όροι στο Βέλιο και Σουηδία, παραδείγματο χάρη, ή αν είναι κάποια πυκνοκατημένη αστική περιοχή ή ύπεθρος. Όλα αυτά, δηλαδή αν συγκρίνουμε την ύπεθρο της Σουηδίας με τη του Βελγίου πάλι έχουμε διαφορές. Ε, η δέσμη των 800 MHz έχει ήδη καθαριστεί και έτοιμη, είναι έτοιμη προς χρήση. Πολύ ωραία. Έχουν εφαρμοστεί σχετικές διατάξεις δηλαδή και λειτουργούν ε, αισίως. Τώρα για την υποζώνη κάτω των 800 μεγαχές για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση ε, αναρωτιέμαι Τι θα κάνουμε, θα το πάρουμε από το, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και θα το δώσουμε στην κινητή τηλεφωνία αυτό το νέο, ε, αυτή τη νέα υποζώνη με τις ε, ραγδαίε τεχνολογικές εξελίξει δεν ξέρουμε ακριβώ ε, σε τι θα μας οδηγήσει αυτό στην ε, Σουηδία. Ε, έχει ήδη εφαρμοστεί η ψηφιακή επίγεια τηλεόραση γιατί δεν υπήρχε, υπήρχε άλλη δυνατότητα. Πολλοί αγόρασαν ε, επίπεδε οθόνε, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε του κανόνε πάλι σε δύο-τρία χρόνια για να του πούμε ότι η νέα σα τηλεόραση ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρειάζεται άλλο αποκωδικοποιητή και άλλο τηλεκοντρόλ. Θα οργιστούν οι καταναλωτέ και δικαίω. Οπότε σας, θα ήθελα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Υπάρχουν πράγματα πρέπει να συνυπολογίσουμε. Στο πακέτο τηλεπικοινωνιών μιλήσαμε και για άλλε λύσει. Να δώσουμε στην κινητή τηλεφωνία τη δέσμη των 800 MHz. Συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε μια απόφαση φέτο και στο, σε δύο χρόνια να αλλάζουμε τη γνώμη μα. Γιατί και η βιομηχανία και οι καταναλωτέ πρέπει να γνωρίζουν τι θα ισχύσει μακροπρόθεσμα. Αυτέ είναι οι βασικέ μου παρατηρήσει. Ε, δηλαδή, η υποζώνη κάτω των 800 πρέπει να παραμείνει στην τηλεοπτική τηλεόραση. Κατά τα άλλα είμαι υπέρ της εναρμόνισης της χρήσης του ραδιοφάσματο. Η κυρία Στήλερ έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Να είστε σύντομοι. Θα είμαι, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με το, τους κυρίους Έλτον και Έγκστρομ. Δηλαδή πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το χρονοδιάγραμμα, για την ψηφιακή μετάβαση. Το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργήθηκε θέμα, παραδείγματο χάρη. Ε, Πώ, εντάξει είναι διαθέσιμη η ζώνη συχνοτήτων, αλλά χρειαζόμαστε ευελιξία, 12 μήνε, 18 μήνε για τη μετάβαση. Ε, να, δεν θέλω να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα αυτό καθε αυτό, αλλά θα είναι ευέλικτο. Αυτό θέλω να μάθω γιατί ε, θα πρέπει να προγραμματίσουν κάποιοι βάση της 12ης ή της 18ης περίοδου. Ε, μπορεί να μας μιλήσει για τη χρονική κλίμακα ε, κάποιος. Η Πρόεδρος ρωτά τον εκπρόσωπο της ευρωπαϊκή Επιτροπής αν έχει κάποια απάντηση να δώσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Συγήτρια για την εξαιρετική σας έκθεση και με τα χαρά θα απαντήσω σύντομα στα θέματα που θίξατε στην τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα όμως συγχρόνως να ε, εντοπίσω ορισμένα θέματα που θίξατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε ήθελε να εξασφαλίσει ότι οι δημόσιες εκπομπές της τηλεοράσεως θα προστατεύονται αποτελεσματικά και θα μπορούν να αναπτύξουν και την ε, ε, τηλεόραση ψηλής πιστότητος και της τελευταίας τεχνολογίας. Ε, τώρα όμως δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία απόφαση χωρίς να, ε, να γνωρίζουμε ποια θα είναι η τεχνολογία σε 5-7 χρόνια. Οπότε ας αφήσουμε ανοιχτό αυτό το θέμα κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία σωστή διαδικασία, να αναθεωρήσουμε το θέμα, να δούμε πώς αναπτύσσονται η ευρυζωνική τεχνολογία και τηλεοπτική τεχνολογία διότι όσον αφορά το ευρυζωνικό σύστημα ε, θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, προχωρούν αποτελεσματικά και να σέβονται τα φάσματα και οι ίδιοι δεσμεύονται να το πράξουν. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και νέα φάσματα και όλες ε, ε, όλες, ε, ό,τι πρόκειται να συμβεί σε 5-7 χρόνια μας είναι ακόμη άγνωστο. Δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα, πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στις μακροπρόθεσμες αλλαγές που μπορεί να συμβούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν καιρό το δέντι όταν θα είμαστε έτοιμοι θα πρέπει να σκεφτεί και να δει πώς η κατάσταση αναπτύσσεται εντωμεταξύ. Επίσης όσον αφορά την εναρμόνιση έχουμε φροντίσει να καλύψουμε τα, τη δέσμη των 300 MHz και να προστατεύσουμε συγχρόνως πέραν της τηλεοράσεως και άλλους δημόσιους χρήστες οι οποίοι χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στα φάσματα. Και τέλος ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που οργάνωσε όλες τις ακροάσεις και τις συζητήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας ε, για ε, τα θέματα. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε μέσω της γραμματείας. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρες, αλλά όσον αφορά τα, την δέσμη των 800 MHz η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε για το 2013 πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά και συνάδει με αυτά που ελέγχθησαν εδώ να υπάρξει αλληλεγγύη προς τις τρίτες χώρες ώστε οι χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν των παρεμβολών των εκπομπών από αυτές τις τρίτες χώρες και να υπάρχει ένας σαφής μηχανισμός για παρέκκληση για το 2015 και για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που υπάρχουν προφανείς λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να είναι ελεύθερες συχνότητες για τους Ολυμπιακούς και ούτω καθεξής θα πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες επενδύσεως και μεταφοράς τεχνολογίες από τους εμπειρογνώμονες διότι χρειάζεται πολύ χρόνος για τη μεταβατική περίοδο της τηλεόρασης και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες αυτές τις προκλήσεις για να διαμορφώσουμε την τελική γνώμη και να πάρουμε απόφαση. Νομίζω ότι τώρα έχει καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμά μας και πρέπει να σας πω ότι με ενθαρρύνει αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ο κόσμος ε, είναι ε, πρέπει να περιμένουμε ώσπου όλος ο κόσμος να είναι έτοιμος και να μην υπάρχουν πλέον εμπόδια. Αφού σας άκουσα λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά και ε, θα διατυπώσουμε από κοινού ορισμένες τροπολογίες. Τώρα, το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ο κύριος Μάντερς και δεδομένου του περιορισμένου χρόνου θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ σύντομοι. Συμφωνείτε κύριε Μάντερς, όχι, εγώ θα φάω όλο το βράδυ. Αν δεν σας πειράζει για την Ανδώρα. No. Uh, just be briefly because it's... Θα ε, είμαι σύντομος γιατί ε, το θέμα μας Ε, είναι ε, να προτείνουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, τη θέση μας. Δεν θέλουμε με αυτό το νέο πρωτόκολλο να επηρεαστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, το νέο πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανδόρας. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Μπορούμε κατόπιν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Σβάπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή δεν είπα τίποτα για τα ε, ραδιοφωνικά φάσματα, σαν σκιώδης εισηγητής ε, θέλω τώρα ε, να παρέμβω σαν εκπρόσωπος της πολιτικής μου ομάδος και να του πω ότι πιστεύω ότι αυτές οι διατάξεις μπορεί να έχουν αρνητικές ε, Επιπτώσει στην εσωτερική αγορά και ε, να του πω ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Ο κύριος Κρίς Βαν Κρίκεν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο γίνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάντερ, τον εισηγητή σας, ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε και εκπώνησε την ε, έκθεση αυτή, όπου με ακρίβεια συνοψίζει την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βασικός στόχος της πρότασής μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο ανάμεσα στην Ένωση και την Ανδόρα θα ε, συνεχίσει απρόσκοπτα, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές βάσει και το πλαίσιο προτύπων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, καταγράφω την ανησυχία σας, το αίτημά σας ότι σε καμία περίπτωση το νέο πρωτόκολλο δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ε, η πρόταση αυτή σχετίζεται βασικά με την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Ε, για το ευρύτερο δωραζήτημα ζήτημα, ενδεχόμενες συνέπειες επί της ενία αγοράς, Δηλαδή, σας παραπέμπω στο πόρισμα των, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ε, του Δεκεμβρίου του 2010 όπου συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση σχετικά με τις ε, δυνατότητες ε, ενσωμάτωσης μικροκρατών συμπεριλαμβανομένης και της Ανδόρας ε, στην ενιαία αγορά. Ε, αυτό προφανώς είναι το ευρύτερο ζήτημα, το είπα, δεν είναι άμεσα θέμα αρμοδιότητός μου, αλλά ε, είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή σας ε, θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία και θα είναι ενήμερη για την έκβαση των σχετικών συζητήσεων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, εμείς σας ευχαριστούμε για την καταθέση τροπολογιών. Η ημερομηνία είναι 2 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι και θα ήθελα να σας πω ότι ε, εφαρμόζεται η διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Είτε θα το εγκρίνει είτε θα το απορρίψει ε, ε, το σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό προβλέπεται στην διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Διακόπτει ο εισηγητής, ο κύριος Μάντες. Συγγνώμη, μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες για την αιτιολογική έκθεση. Δηλαδή θα πούμε ναι ή όχι, θα συμφωνήσουμε ή δεν θα συμφωνήσουμε για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα επιτρέπετε. Ήταν ένας αστεϊσμός του κ. Πρόεδρος, ε, ξέχασα να σας ε, να αναφέρω την πρόταση υποβολής, ε, τη, συγγνώμη, την προθεσμία τροπολογιών για το προηγούμενο θέμα. Στις 4 Μαρτίου ήταν, στις 12, για το προηγούμενο σημείο ήταν αυτό. Και κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω, κυρία Στήλερ, κάνατε μία ερώτηση. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του 2013 με κάποιες εξαιρέσεις όταν είναι ανέφικτο, αδύνατον να ακολουθηθεί ε, πιστά το χρονοδιάγραμμα, όταν το δικαιολογούν ε, οι περιστάσεις. Um, yes. Now we go of Τώρα, παρουσίαση από την ομάδα εργασία ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ε, gracias, Presidenta. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, εμείς έχουμε μοιράσει την παρουσίαση και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το παρακολουθήσουν στην συνθήκη. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτήν την ε, έκθεση. Όπως ήδη συζητήθηκε ευρύτατα σε αυτήν την Επιτροπή, η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί ένα μέσο με τεράστια δυναμική για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς και την ενίσχυση του, της ανταγωνιστικότητάς μας και εμείς αυτό το πλεονέκτημα μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να σας αναλύσω το σενάριο του ηλεκτρονικού εμπορίου σήμερα στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια ξεπερασμένη νομοθεσία και τεχνολογική καθυστέρηση. Δεν έχουμε, κανένα, δεν έχουμε ελάχιστους ελεγκτικούς οργανισμούς, έχουμε έλλειψη διαφάνειας και αυτό συνδέεται και με την ανασφάλεια και την έλλειψη εμπιστοσύνης του καταναλωτή. Αυτό το σενάριο οδηγεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη σε ανεπαρκή ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Πού θέλουμε όμως να φτάσουμε, τι θέλουμε εμείς ως σενάριο. Εμείς θέλουμε σαφήνεια, ρυθμιστική σαφήνεια και οργανισμούς ελέγχου που να εγγυούνται καλές πρακτικές. Θέλουμε εμείς κίνητρα για τους πολιτές και για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέλουμε ενιαίο ΦΠΑ. Θέλουμε εγγύηση για τους καταναλωτές και ξεπέρασμα των τεχνικών συνόρων με συνδέσεις υψηλής ποιότητας. Έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε μια αγορά με πάνω από 500 εκατομμύρια χρηστών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να κάνουμε μία ανασκόπηση των τοποθετήσεών μας και να βρούμε νέους δρόμους. Επιτρέψτε μου μετά από αυτήν την εισαγωγή να σας παρουσιάσω το σχέδιο γύρω από το οποίο εργαζόμαστε. Πρόκειται για μία πρόταση που μπορεί να πάρει τη μέση οδό μεταξύ των δύο σεναρίων που σας παρουσίασα. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σήμα, ένα ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας το οποίο θα δημιουργούσε, θα έδινε και τις απαραίτητες εγγύησεις στον καταναλωτή για τις συναλλαγές του στο ίντερνετ υπό το δίκτυο EUR. Θα δίνεται εγγύηση ότι όλες οι συναλλαγές του θα καλύπτονται από την νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα πληροφορεί. Πρόκειται λοιπόν για υποδομή πληροφόρησης για τη δημιουργία εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό το σήμα θα, είχε, θα πληροφορούν τον χρήστη αναλυτικά για όλα τα ζητήματα σχετικά με τις συναλλαγές που θέλει να πραγματοποιήσει και θα, με τελικό στόχο τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Καταναλωτές, ε, θεσμικά όργανα, χρήστες όλων των ειδών θα καλυπτόντουσαν από μία ενιαία οδηγία δικαιωμάτων του καταναλωτή, μία ενιαία ε, νομοθεσία προστασίας δεδομένων και απόλυτη πληροφόρηση για το προϊόν και για τον πολιτή με ασφαλείς δυνατότητες πληρωμής και με τιμές ανταγωνιστικές. Υπάρχουν όμως αντιρρήσεις σε αυτό το σχέδιο. Οι καταναλωτές έχουν μία ανικανοποίητη επιθυμία. Θέλει να, να αγοράσει ο καταναλωτής αλλά δεν έχει ασφάλεια. Οι ενώσεις και οι χρήστες και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα. Ασφάλεια και εμπιστοσύνη, η αύξηση των εμπορικών πανευρωπαϊκών συναλλαγών θέλουν να έχουν κοινή φορολόγηση και ενιαίους λογιστικούς κανόνες, ελεύθερο ανταγωνισμό με μια καλύτερη εποπτεία της αγοράς και μεγαλύτερο ή ενδυνάμει αγορά μέσα από την ασφάλεια και την διαφάνεια. Βασική λοιπόν αντίρρηση η έλλειψη εμπιστοσύνη και αυτό λόγω της πολυπλοκότητας και ανισότητας της νομοθεσίας για τα υπάρχοντα κενά και την έλλειψη των, της πολιτικής βούλησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να εξεταστούν και να ληφθούν τα απαραίτητε μεταρρυθμίσεις. Οι ενώσεις επίσης θα κέρδιζαν θα, μεγάλωνε η αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές θα είχαμε μεγαλύτερο έλεγχο της πειρατείας και των προϊόντων που βλάπτουν τη δημόσια υγεία. Κάτι τέτοιο θα ε, βοηθούσε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας εσωτερικής αγοράς από τη θεσμική πλευρά που εκπροσωπούμε πολλοί από τους παρόντες ε, σε αυτή την αίθουσα είναι να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τις διάφορες οργανώσεις και ενώσεις. Πρέπει να συμμετέχουν λοιπόν τα stakeholders σε αυτό, σε αυτό το σχέδιο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σχέδιο. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την ενιαία αγορά σε πραγματικότητα. Υπάρχει μία βούληση, σαφέστατη βούληση, αλλά και μία πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώσει την ψηφιακή αγορά. Και εδώ σε αυτή την παρουσίαση έχετε μερικά παραδείγματα. Πρέπει να έχουμε το όραμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν αυτό το μέσο θα μπορούσε να μας βοηθήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο να ξεπεράσουμε την κρίση να βγούμε από τις οικονομικές δυσκολίες. Σε αυτή τη φάση κρίσης δεν θα πρέπει εμείς να εξοικονομήσουμε προσπάθειες σε ό,τι θα μπορούσε να μας επιτρέψει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Ευθύνη μας είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως την αγορά των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών. Είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται καινοτομία, απλούστευση, επικοινωνία και εγγύηση. Θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την Trust που αναφέραμε προηγουμένως και θέλουμε να πετύχουμε εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτές είναι οι ιδέες μου για το θέμα. Και με αυτό το στόχο και υπ' αυτήν την οπτική θέλω να εξετάσουμε την ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μια ανοιχτή ομάδα εργασίας, διότι η παρουσίαση που κάνω σήμερα εδώ παρουσιάζει τις δικές μου προσωπικές ιδέες για το θέμα. Αποτελεί απλά και μόνο μια φετηρία, μια πρόταση. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι οι συνάδελφοί μου, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν και οι εκπρόσωποι των stakeholders θα μπορέσουν να συμμετέχουν για να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση. Στην αρχή της παρουσίασης ανέφερα ποια είναι η τωρινή κατάσταση, κατάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε και που χρειάζεται αδιαμφισβήτητα μία ε, νέα μία αναδιοργάνωση, ένα νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της ομάδας εργασίας ε, και ευτυχώ υπάρχει ένα μέλος της ομάδας εργασίας ε, παρόν. Θα ήθελα πριν σας δώσω το λόγο να τονίσω τη σημασία που έχει η ομάδα εργασίας αυτή για το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες για να τονώσουμε την οικονομία της Ευρώπης, την εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα. Ε, ουσιαστικά θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα εργαλείο για να ε, εξέλθουμε από την κρίση, αλλά θα πρέπει να επικαιροποιηθεί αυτό το εργαλείο, ε, διότι η κοινωνία του 21ου αιώνα είναι ψηφιακή. Ο κύριος Κορίντε Κάμπος μας έχει... θα πάρει το λόγο, είναι μέλος ομάδας εργασίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παύλο Άριας. Ήταν εξαιρετικά ποιοτική η παρουσίασή του και έδειξε μεγάλη επιμονή για να προωθήσει ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η παρουσίασή του. Θα ήθελα ήθελα, επειδή δεν τη γνώριζα εκ των προτέρων, να εκφράσω τρεις ε, αμφιβολίες ή τρία σημεία προς προβληματισμό, προς ε, ε, ε, μελλοντική συζήτηση. Το πρώτο σημείο σχετίζεται με τα προβλήματα, τις διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν όταν γίνεται προσφυγή για την εγγύηση, πώς να το πω, όταν υπάρχει μια ιονή παραβίαση του νόμου, επειδή κάποιοι θέλουν να επωφεληθούν ε, από τα προνόμια χωρίς όμως να υποστούν το κόστος και τους περιορισμούς ε, Αυτό θα πρέπει να το δούμε, αυτό το σημείο πρέπει να το δούμε πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ο καταναλωτής ε, θα φορτωθεί το λειτουργικό κόστος ε, του συστήματος. Προφανέστατα θα υπάρχει λειτουργικό κόστος. Ποιος θα πληρώσει ο καταναλωτής, έμεσα βέβαια, δηλαδή οι ε, κατασκευαστές και οι πολίτες ε, που θα ε, ανταγωνίζονται μεταξύ τους μπορεί ή μάλλον όχι μπορεί, σίγουρα θα θέλουν να απαλλαγούν από αυτό το κόστος και θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Κατόπιν, μια πιο συγκεκριμένη σύσταση από πλευράς μου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πολετομιακή ομάδα εργασίας. Ε, ο κύριος Αρίας ε, εξ αρχής ε, επέμεινε για τη σύνθεση της ομάδας, δηλαδή να συμμετάσχουν βουλευτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι stakeholders, από τη βιομηχανία, από τις επιχειρήσεις κτλ. Ήδη λοιπόν ε, ε, στην πρώτη φάση της διαδικασίας σαν οι εμπλεκόμενοι φορείς και εγώ δεν συμφωνώ διότι μπορεί, ε, επειδή οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ίδια συμφέροντα δέχεται να παραμορφωθεί ο ορισμός της βασικής έννοιας. Μην ξεχνάτε ότι εκείνοι βλέπουν το πρόβλημα από το δικό τους οπτικό πρίσμα ε, το οποίο δεν είναι το ίδιο με αυτό των καταναλωτών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε εμείς οι βουλευτές. Ε, οπότε δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι πρέπει να διευρυνθεί ε, ήδη από τα αρχικά στάδια τη διαδικασία η σύνθεση ομάδα σε όλου του εμπλεκόμενου φορεί. νομίζω ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθούν τα θεσμικά όργανα και κατόπιν αν υπάρχει ε, κάποια ε, συγκεκριμένη ε, πρόταση τότε να συμμετάσχουν ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς για να μπορέσουμε και εμείς να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αυτά είχα να σχολιάσω και ευχαριστώ τον συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Η κυρία Στήλερ και ο κύριος Σφάπ έχουν ζητήσει το λόγο. Κυρία Στήλερ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για την εξαιρετική παρουσίαση. Ε, είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία ε, και θα ήθελα να σχολιάσω μόνο ένα θέμα. Μιλήσαμε για το συμβατικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Οικονομικών Υποθέσεων και στη δική μας Επιτροπή. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για αυτό το θέμα. Δηλαδή επηρεάζει αυτό άμεσα ε, το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, όταν εξετάζουμε το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ε, συζητούμε με τους εμπλεκόμενους φορείς ε, για το ΕΒΡΕ 3 και 5 και συζητούμε τα πρότυπα, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξίζει να αναλάβει κανείς αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνήθως συζητάμε μόνο ε, στο Κοινοβούλιο για προτάσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ εδώ πρόκειται για μία πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου και ε, έχω δει την πρόταση του συναδέλφου Αρίας την οποία βρίσκω την, ε, ως πολύ ενδιαφέρουσα διότι όπως είπε η κυρία Στάιλερ συνδέεται με άλλες προτάσεις για την εναρμόνιση της εσωτερικής εξωτερικής αγοράς ή θέματα που αναφέρονται στο Single Market Act ε, σχετικά με το επίπεδο του ΦΠΑ και θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι θετική. Ε, μάλιστα ε, η αντίθεση με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσπαθούν κάτι να πουλήσουν και πρέπει να αποφασίσουν για ένα θέμα αν θα ασχοληθούν με το κοινοτικό επίπεδο ή το εθνικό επίπεδο το οποίο ίσως είναι χαμηλότερο από το κοινοτικό. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει σχετικά με το θέμα αυτό είναι αν τα θέματα αυτά έχουν σχέση με ε, το, τα ντομέν ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εγώ θα ήθελα να πω ότι έχω ένα δικό μου τέτοιο ντομέν μία ιστοσελίδα και θα ήθελα να ξέρω εάν και άλλοι βρίσκονται στην ίδια θέση γενικώ όμως θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με την πρόταση αυτή Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ Κύριε Αρία, θέλετε να διατυπώσετε το πρόγραμμά σας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Εγώ πιστεύω όλα αυτά, ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εδώ είναι αυτά που θα θέλαμε να συζητήσουμε μέσα στην ομάδα εργασίας. Και ο στόχος μου σήμερα ήταν να σας καλέσω σε σκέψη γύρω από το θέμα. και οι τοποθετήσεις σας ε, επιβεβαιώνουν ε, τις προθέσεις μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράσει ο καθένας τις σκέψεις του για την αρχική πρόταση που αποτελεί και ένα πρώτο βήμα προς το στόχο. Φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου το απόγευμα από τις 3 και έπειτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.